Καλημέρα σα. Πάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης να βελτιώσουμε την ποιότητα της δαπάνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζει σήμερα τη θέση του για τρία ντοσιέ υψής της σημασίας και που θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ε, δαπάνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2013 και αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Μετά από πρόταση του συναδέλφου Χατζημαρκάκη, η Επιτροπή μας αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2010 να οργανώσουμε ε, αυτή την ανταλλαγή απόψεων και με εμβάθυνση για την βελτίωση της ποιότητας των δαπανών. Και αυτό ε, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου του 2010, για την, του 2010 συγγνώμη, για την βελτίωση της ποιότητας των δαπανών όπως και το αντίστοιχο κείμενο της Κομισιόν. Όλα αυτά είναι σημαντικά μηνύματα για όλες μας για όλα μας τα θεσμικά όργανα και μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε άποψη για το πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών. Ευχαριστώ τους παρόντες, όλους όσους θα μιλήσουν και θα ξεκινήσουμε από τον συνάδελφο Χατζημαρκάκη που είναι εισηγητής και θα μας αναφέρει σχετικά. Θυμόμαστε τον, τον πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου που έθεσε το θέμα του προϋπολογισμού Θυμόμαστε επίσης την κυρία Θάτσερ πριν μερικά χρόνια που είπε θέλω τα χρήματά μου πίσω. Τώρα λέει ο κύριος Κάμερον δεν θα δώσω άλλα χρήματα, δεν θα δώσω πλέον χρήματα διότι έρχεται αρκετά χρήματα και δεν ξέρω αν τα ξοδεύεται με τον κατάλληλο τρόπο. Ε, δεν είμαι τόσο βέβαιος για το πρώτο σημείο. Νομίζω ότι ε, Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξοδέψει κανείς ε, χρήματα, αλλά μετά τη διαδικασία της αλλαγής και το, την ε, το πώς ξοδεύονται τα χρήματα, κυρίως τα κράτη-μέλη, ως προς την ποιότητα των δαπανών, Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι θα έπρεπε να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που συνέβαλαν στη διαδικασία της απαλλαγής όπου μπορέσαμε να διευκρινίσουμε ορισμένα στοιχεία των δαπανών όπου μπορούσαμε να αναλύσουμε ε, πού μπορούν να βελτιωθούν οι δαπάνες κυρίως από τα κράτη-μέλη αλλά δεν ε, απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν πρέπει να συνεχίσουμε γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ μαζί για αυτήν την ακρόαση και στον David Bostock ευγνώμων από το ελεγκτικό συνέδριο εδώ και μερικά χρόνια ε, και είναι από το ίδιο κράτος μέλος των δύο πρωθυπουργών που ανέφερα. Ωστόσο, μπορούμε ακόμη να πούμε ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι αυτά τα κράτη-μέλη και ο David Boston το ξέρει καλά ε, το οποίο, τα οποία φωνάζουν αυτά που θέλουν να αλλάξουν είναι αυτοί που έχουν ε, προβλήματα στις δαπάνες τους ε, στο, στο δικό τους το σπίτι. Όλα τα προγράμματα της Αγγλίας διεκόπησαν το έτος 2010, όπως ίσως γνωρίζετε. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών, αυτό είναι μεγάλη προτεραιότητα, όχι μόνο για την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, αλλά και για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προετοιμάζουμε τη θέση μας σε τρεις σημαντικούς φακέλους ε, και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να αφαιρθώ πρώτα απ' όλα στην αναθεώρηση ε, του δημοσιονομικού κανονισμού ε, και δεύτερο τον δεύτερο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2013 και τρίτον την ανασκόπηση ε, του ε, προϋπολογισμού και κάθε ένας από αυτών τους φακέλους μας δίνει ευκαιρίες ε, για να εντοπίσουμε τις αδυναμίες που διαπίστωσε το συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει δύο έγγραφα για την βελτίωση των δαπανών στα όργανα του Ευρωπαϊκή Ένωσης και είναι μια πηγή έμπνευσή για τη βελτίωση των δαπανών της χρήσης των κονδυλίων. Χαίρομαι που ήρθε εδώ ε, το ελεγκτικό συνέδριο για να μας πει ε, πώς θα ε, βελτιώσουμε σχετικά με την γνώμη 1-2011 και επίσης για τις κινδύνους και προκλήσεις και έχουμε επίσης συναδέλφους από άλλες επιτροπές που είναι πάρα πολύ σημαντικές σε σχέση με το θέμα αυτό η κυρία Ιούτα Χόκα από την Σούρε ε, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τις ε, κινδύνους και προκλήσεις. Κυρία Περβόνς ε, Περές που είναι επικεφαλής της Επιτροπής Κοινωνικών Αποθέσεων και Απασχόλησης, μια από τις επιτροπέ που ξοδεύει πολλά. Κυρία Μπαλτσάνη που είναι η για τον προϋπολογισμό 2012, Ευρή Ούσδος που είναι συντονίστρια για την Επιτροπή Αλίας. Αλλά τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον David Bostock και ίσως να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Μπόστορ και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή Ελεγχού Προπολογισμού για την σημερινή πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να κάνω λόγο για την ποιότητα στι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κάνοντα αυτό, θα αναφερθώ πράγματι στην άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπαριθμών 1 2010 με τίτλο «Βελτιώνοντας την ε, οικονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ε, και την γνωμοδότηση 6-2010 για τις προτινόμενες αλλαγές για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Καμιά φορά θεωρείται ότι το μόνο σημαντικό θέμα για την ποιότητα των ευρωπαϊκών δαπανών ήταν πώς να αρθούν τα σφάλματα, θέματα τυπικότητας και κανονιστικά θέματα. Υπάρχουν όμως και άλλες συνιστώσεις. Η οικονομία, αποτελεσματικότητα, στην υψηλή ποιότητα. Δεν θα έχουμε υψηλή ποιότητα στις δαπάνες μέχρι ότου βελτιωθεί η επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το τακτό και για το ε, εντάξει των δαπανών. Ξεκινώντας να θέσω κάποια θέματα από τη νομοδότηση υπαριθμών 1 του 2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρώτον, το εντάξει και το δεν είναι καλός. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολλές φορές περίπλοκους κανονισμούς και κανόνες και πολλές φορές είναι αντικείμενο επίμαχων ελεγκτικών συστημάτων. Όμως αυτά τα συστήματα έχουν έναν ανάμεικτο βαθμό επιτυχίας διασφαλίζοντας ότι θα γίνονται σεβαστά αυτά τα σχέδια επιχειρηματολογία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε τέτοιε περιπτώσει μπορούν να υπάρξουν επανορθώσει, διορθώσει. Όμω ε, δεν μπορεί να διορθωθούν ατομικά σφάλματα και εν πάση περιπτώσει παίρνει και πολλά χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο, αν είναι κάτι τέτοιο δυνατόν. Δεύτερον, Υπάρχουν προγράμματα δαπανών όπου η πρόσθετη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προφανή, δεν είναι πρόδειλη. Για παράδειγμα, αυτό ήταν κύριο έβριμα στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου για το 2009 για τι δαπάνε για τη δημόσια υγεία. Τρίτο υπάρχει επανειλημμένη αποτυχία να θεσπιστεί και να καθιερωθεί πώς οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επιτύχουν τα αναμενόμενα, τους αναμενόμενους στόχους, τους προσδοχόμενους στόχους. Γνωρίζουμε ότι αυτό για παράδειγμα στις εκθέσεις μας για τα δίκτυα ε, βέλτιστης επίδοσης ε, για την συνοχή για το 2008 και τις ε, μας για την, την έκθεσή μας για την ευφύ χρήση ενεργειακών πόρων του ίδιου έτους. Τέταρτον, σε κάποιες περιπτώσεις πληρωμές από τον προϋπολογισμό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν προσαρμογέ με κριτήρια τα οποία δεν μπορούν άμεσα να επαληθευθούν. Η δική μα έκθεση υπαριθμών 8-2008 βρήκε ότι η διασταυρούμενη συμμόρφωση για τη γεωργία δεν μπορεί να ελεγχθεί πάντα από τους ελεγκτές. Πέμπτον, και ίσως το πιο σύνηθε παράπονο τα προγράμματα έχουν ελλείψεις και λύματα όσον αφορά την εποπτεία και την αξιολόγηση. Είναι συχνά δύσκολο να βρει κανείς ε, ποιες είναι οι βέλτιστες δηλώσεις για αυτά, για το πόσο έχουν κοστίσει κάποια προγράμματα, ποιος επομίστηκε το κόστος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, οι εποφελούμενοι και τι έχει επιτευχθεί με όλα αυτά. Όλα αυτά είναι αρκετά θλιβερά, αλλά η γνωμοδότηση υπαριθμών 1 2010 δεν ήταν μόνο μια άσκηση σε ζωφερά θέματα και απεσιοδοξία. Επεσήμανε κάποιου τομεί ε, το ελεγκτικό συνέδριο που κάποια πρόοδο θα μπορούσε να επιτευχθεί και κάποιε λύσει που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, να υιοθετηθούν. Ένα θέμα τη γνωμοδότηση είναι ότι η ποιότητα πρέπει να ενταχθεί ευθύ εξ αρχή ε, στι δράσει τα προγράμματα δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι ανανεώνονται χωρίς σωστή αξιολόγηση με βάση κάποιες μικροαλλαγές στα ποσά αντί να υπάρχει μια εκβάθρον επαναξιολόγηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημειώσαμε για παράδειγμα στην έκθεσή μας του 2008 για την χρήση με φύ τρόπο των ενεργειακών πόρων, όπου σε διάφορα υποπρογράμματα που επανειλημμένα ανανεώθηκαν, χωρίς να υπάρχει έκθεση αξιολόγησης για τις προηγούμενες δαπάνες για αυτά προηγούμενα. Η γνωμοδότησή μας λοιπόν υπαριθμών 1-2010 είναι ένα εγχείρημα για τις δράσεις που μπορούν να αναλυθούν προτού, αναλυθούν τέτοια προτού δομολογηθούν τέτοια προγράμματα. Επισημαίνει το ελεγκτικό συνέδριο στη μελέτη επισημα... Ε, αξιολόγησης επιπτώσεων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει με μια σε βάθος εξέταση του κόστους και των ωφελιών μιας τέτοιας δράσης. Μια σωστή αξιολόγηση και ε, αξιολόγηση και των εναλλακτικών λύσεων. Καμιά φορά καλύτερο είναι να κάνει κανείς κάτι παραπάνω, καμιά φορά κάτι παραπα... παρακάτω, κάτι λιγότερο, καμιά φορά και τίποτα. Είναι σημαντικό θέμα το θέμα της απλούστευσης. Απλούστευση κανονισμών και κανόνων που <clears throat> πιθανότατα προχώρησε περισσότερο στον τομέα της γεωργίας από ό,τι σε άλλους τομείς. Είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς το συμπέρασμα ότι αυτή η απλούστευση συνεισέφερε σημαντικά σε χαμηλότερα ποσοστά σφάλματος σε σχέση με τα όσα είχαμε βρει στα τελευταία χρόνια για τις δαπάνες της ΚΑΠ. Εν τέλει, πρότεινε το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εκβάθρον αξιολόγηση όσον αφορά τις επιδόσεις και τα ωφέλη των αποδεκτών σε σχέση με το output και input. Τώρα, στρέφομαι στον δημοσιονομικό κανονισμό που προκάλεσε πολλή δουλειά και στο, στο ε, ε, κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως και προηγούμενα σε σχέση και με το ίδιο το Ελληνικό Συνέδριο. Μία προειδοποίηση. Δεν θα πρέπει εδώ να έχουμε μόνο διεύρυνση του, του πλαισίου για την καλύτερη ποιότητα. Χρειάζεται τομεακή νομοθεσία. Καλύτερη τομεακή νομοθεσία επιπλέον και όχι μόνο γενικά μέτρα. Είπε αρκετά το Ελληνικό συνέδριο για αυτό το δημοσιονομικό κανονισμό στην νομοδότηση 6-2010 για παράδειγμα κυρίως. Και αν επιτρέπετε εμείς σήμερα θα μπορέσουμε να παραστούμε και μέχρι και το απόγευμα αν συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα προχωρήσω σε τρεις άξονες που είναι σημαντικοί. Η έλεγχη, οι λογαριασμοί και το ανεκτό σφάλμα, ανεκτό επίπεδο σφάλματος. Εξωτερική έλεγχη. Έλεγχη των δαπανών είναι μια πολύ προκλητική δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελεγκτές μας πρέπει να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια πρέπει να εργάζονται με βάση ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Είναι μια δουλειά που απαιτεί μεγάλη ελαστικότητα και συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι και μεταξύ τρίτων εμπλεκομένων ε, πλευρών. Είναι σημαντικό ο δημοσιονομικός κανονισμός να μην παρακολεί αυτό το έργο. Δυστυχώς Κάποιες από τις προτάσεις για τους εξωτερικούς ελέγχους που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχαν παρακολλήσει αυτό το έργο αλλαγές, εισάγοντας αλλαγές που θα περιόριζαν το έργο αυτό. Γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο στράφηκε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να απορριφθούν πολλά στοιχεία προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τέτοιους ελέγχους. Οι λόγοι και οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην νομοδότησή μας 6-2010. Δεύτερον, οι λογαριασμοί. Ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα τελευταία έξι χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιτυχία υλοποίησε τις προδιαγραφές για τους δημόσιους λογαριασμούς. Εξεπλάγημεν γι' αυτό στο Λουξεμβούργο να δούμε ότι το σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να οπισθοχωρεί από αυτό το πλαίσιο και να... αυτό να μην είναι θετικό από τις συζητήσεις όσον αφορά την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τώρα έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι γνωρίζω, ένα νέο, μια νέα πρόταση που καθορίζει ένα πιο σωστό πλαίσιο για τους λογαριασμούς αυτούς. Και ελπίζω ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια γραμμή θα ακολουθήσει και στις συζητήσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτον και τελευταίο, να πω δύο λόγια για το ανεκτό επίπεδο σφάλματος. Το ελεκτικό συνέδριο επί ε, δια Μακρόν είχε ασχοληθεί για το κόστος ε, του διοικητικού βάρους που πολλές φορές είναι δυσανάλογο σε σχέση με τα ωφέλη που δίνονται, που απορρέουν και θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πώ είναι δυνατόν όχι μόνο να είναι αποτελεσματικά τα συστήματα ελέγχου αλλά να είναι αποτελεσματικά και όσον αφορά τι δαπάνε ε, που θα συνεπάγονται. Υπέβαλε προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα ανεκτό επίπεδο σφάλματο ε, στι προτάσει τη για τον δημοσιονομικό κανονισμό και από ό,τι γνωρίζω οι εισηγητέ σα βλέπουν κάποιο κίνδυνο αυτέ οι προτάσει ε, να θεωρηθούν ως αλλαγή του πλαισίου και σε σχέση με τις ε, απαιτήσει ε, που τίθενται στις ε, δημοσιονομικές ελεγκτικές αρχές και κατανοώ την ανησυχία των εισηγητών. Επεσήμανε λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο ότι το πιθανό επίπεδο σφάλματος και το πιθανό κόστος των συστημάτων ελέγχου είναι πράγματα που πρέπει να εξεταστούν όταν νέες προτάσεις υποβληθούν και όχι κάτι να εξεταστεί όταν θα εξετάσει την χωρίση απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύτερο θα είναι αυτό να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο στον δημοσιονομικό κανονισμό, ώστε να υπάρξει σωστή αξιολόγηση του κόστους κόστους εφαρμογής και υλοποίησης, καλύτερη αξιολόγηση δηλαδή των κινδύνων των πραγμάτων που παρεκκλίνουν και δεν πάνε καλά, όταν οι προτάσεις υποβάλλονται αντί να υπάρξουν νέε απαιτήσει εκ των υστέρων που θα επιβάλλονται στι ε, αρχέ χωρίσει τη απαλλαγή, Αυτά για τον υποσυνομικό κανονισμό. Πρέπει να ολοκληρώσω λέγοντας δύο λόγια για το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται αυτή η συνεδρίαση παρότι ίσω μάλλον επαναλαμβάνω τα όσα είπε ο κύριο Χατζημαρκάκη πιο πριν. Η οικονομική κατάσταση σίγουρα έγινε δυσκολότερη από τότε που είχαμε την γνωμοδότηση του 2010. Και όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκοτία, ε, Ουαλία, ε, Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση είναι χειρότερη από τότε. Πολλές, ε, πολλά κράτη έχουν προβλήματα με το ευρώ. Πρέπει να δαπανά σωστά τα κονδύλια που έχει στη διάθεσή τη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το δικαιολογεί αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσβλέπω στο να ακούσω τι απόψει των άλλων ομιλητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, σα ευχαριστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον David Μπόστοκ για την παρουσίασή του και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Χάουαρντ ε, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Η κυρία Χάουκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Πρέπει όμως ε, εκ προημίου αμέσως να πω ότι η Επιτροπή έχει μια περιορισμένη εντολή Φυσικά δεν επιτρέπεται να αναμειγνιόμαστε στι στις αρμοδιότητες των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών όσον αφορά για παράδειγμα την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού προσπαθώντας να δώσουμε εμείς κάποιους κανόνες ή κανονισμού. Συζητήσαμε λοιπόν τι είναι αυτά που αφορούν την συμφωνία για την υλοποίηση του προϋπολογισμού μα συνολικά, όχι μόνο για τα μεγάλα κονδύλια, αλλά και για τα μικρότερα κονδύλια. Και έχουμε διαφορετικές, ας διαφορετικά συστήματα διαχείρισης κάποια ταμεία, κάποια κονδύλια δαπανώνται από τα κράτη-μέλη. Κάποια άλλα, τα μικρότερα κυρίως, κεντροποιημένα διαχειρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς συζητήσαμε για αυτά τα θέματα. Ποιες βελτιώσεις ε, μπορούν να υπέρθουν. Το μόνο που είχαμε ως πρόταση, ως στοιχείο, ήταν η έκθεση ακριβώς του ελεγκτικού συνεδρίου. Μας είχαν υποσχεθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θα είχαμε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υπεβάλλω το, για την απλούστευση. Όμως, αυτή η ανακοίνωση μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί, δεν έφτασε στα χέρια μας και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καν αυτή η γνωμοδότηση, η ανακοίνωση. Ο εισηγητής μας τελευταία φορά στις 30 Μαρτίου με το γραφείο του Επιτρόπου Σέμετα συναντήθηκε και προσπάθησε κάποια πράγματα να πάρει επειδή θέλαμε στις δικές μας, στα δικά μας συμπεράσματα της τελικής μας έκθεσης να συμπεριλάβουμε αυτά τα στοιχεία. Τώρα αυτό θα απουσιάζει δυστυχώς πρέπει να πω γιατί δεν είχαμε, δεν έχουμε καμιά δυνατότητα να πάρουμε τέτοια στοιχεία. Θα μπορούσαμε να πούμε δημοσιονομικός κανονισμός καταρχήν. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για την απλούστευση. Αλλά και πάλι σε αυτό το σημείο δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Θα παραμείνουν λοιπόν τα πράγματα έτσι. Δηλαδή ότι απευθύνουμε έκκληση και ζητούμε, απαιτούμε για όλα τα ταμεία και κονδύλια με κοινέ αρχές να διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά. Και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει οικονομικότητα, σωστή διαχείριση και αποτελεσματικότητα. Σε αυτά δίνουμε μεγάλη αξία. Όμως για διάφορα μέσα ή διάφορους ε, τομείς πολιτικής ε, δεν είναι δυνατόν να, να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ε, ανάμειξη εμβάθυνση. Και το λέω αυτό ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα όταν θα έχει συμφωνηθεί και ψηφιστεί η έκθεση 25-26 Μαρτίου αντίστοιχα. Τότε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ξαναδούμε τι πρέπει να γίνει όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, τον δημοσιονομικό κανονισμό. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι στα μεγάλα ταμεία όπου εκείνο που θέλουμε είναι στα κράτη-μέλη πραγματικά πολλά κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να μπορούν να δαπανώνται, σύμφωνα με τους δικούς μας στόχους και τη δική μας ε, άποψη για τη χρήση, να υλοποιούνται αυτά όλα. Και ότι έχουμε εκεί ένα μέρος ε, των κονδυλίων που διατίθενται στα ταμεία, που χρησιμοποιείται ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν μια, ας το πω έτσι, κατεύθυνση και βοήθεια για την better governance, την σωστότερη, καλύτερη διαχείριση και για ένα χρονικό διάστημα βοήθεια για την στελέχωση, για τα στελέχη, manpower. Γιατί βλέπω ότι πολύ συχνά, γι' αυτόν τον λόγο, οι απόψεις που έχουμε αναπτύξει και εν τω μεταξύ έχουμε και μια τρίτη δημοσιονομική πρόβλεψη εδώ, ένα τρίτο πλαίσιο το οποίο αναπτύσσουμε για δημοσιονομικές προοπτικές και κάθε φορά είχαμε απόψεις και ιδέες και κάθε φορά όταν είχαμε μεταρρύθμιση του μέσου αυτού για την περιφερειακή πολιτική και τη διαθωτική πολιτική κάθε φορά όταν είχαμε τα θέματα της γεωργικής πολιτικής θέλαμε και θέλουμε να είναι τα πράγματα πιο αποτελεσματικά και πιο σωστά και κάθε φορά βλέπουμε ότι πολλές φορές σε διάφορου τομεί υπάρχουν ελλείψεις, ελληματικές καταστάσεις. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς θα έπρεπε ίσως σε σχέση με τις επιδόσεις των κρατών μελών, ας το πω έτσι, να μην υπερεκτιμούμε τα πράγματα. Υπερεκτιμούμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη, και δεν εννοώ τα νέα εδώ, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη, δεν εννοώ τα νέα, με συγχωρείτε, τα νέα κράτη-μέλη λέει η ομιλήτρια, ότι δεν υπάρχει εκεί η διαχείριση που επιθυμούμε, ώστε περιφερειακά, τοπικά, όλα να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να πετύχουμε τους στόχους μας, ενώ και άλλα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν ε, είναι, είναι κάτι το οποίο θα εντασσόταν στην έκθεσή μας, διότι δεν βρίσκεται αυτό στην εντολή μας. Και δεν είναι αυτό κάτι που είναι επίσημη άποψη, είναι ιδιωτική άποψη, κατηδίαν που έχουμε και προσπαθώ με τους αρμόδιους για την γεωργία και τους υπεύθυνους ε, για την περιφερειακή πολιτική από εμάς στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Ευρωβουλής προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε και έτσι να προβληματιστούμε τι πρέπει να γίνει στο μέλλον ώστε όταν θα έρθει η ώρα της πραγματικής νομοθεσίας για τα διαθροτικά ταμεία για την, τον επόμενο γύρο της αναθεώρησης της γεωργικής της αγροτικής πολιτικής να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο προς αυτές τις κατευθύνσεις. Αυτά ήθελα να πω για αυτό το θέμα και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε στον επόμενο γύρο δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά όχι μόνο για τα μεγάλα ταμεία, όπου έχουμε μεγάλη μεγέθυνση, ας το πω έτσι, ε, θέμα μεγέθυνσης της επίτευξης των στόχων μας, αλλά και για τα μικρότερα ταμεία, όταν πρόκειται για καινοτομία ή έρευνα, για παράδειγμα, ή για την κατεύθυνση εκείνων που ασχολούνται με την έρευνα και την ε, ανάπτυξη ή με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουμε πραγματικά δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες καινοτομίας και χρειαζόμαστε τότε απλούστευση. Και για αυτούς όλους τους λόγους ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο εδώ. Αλλά και γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο λόγω ε, έλλειψης εντολής και δεν θέλω εδώ να υπάρξει αντίθετη άποψη από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Χάουκ. Τώρα έχει το λόγο η συνάδελφος Μπερές, πρόεδρος της Οπιτρεπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για την πρόσκληση σας προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που διαχειρίζεται ορισμένα προγράμματα και κανονισμούς που είναι χρήσιμοι για την εφαρμογή ορισμένων στρατηγικών που απορροφούν επίσης ένα μέρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θεωρώ κατά συνέπεια ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στη συζήτηση κυρίως στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 για την ποιότητα της δημόσιας δαπάνης. Γι' αυτό μας καλέσατε. Ε, και πάντοτε με τους συνομιλητές μας έχουμε ένα τεράστιο ερώτημα. Πώς αξιολογούμε την ποιότητα. Ποια είναι η ποιότητα, το χαμόγελο των δικαιούχων που έχουν βγει από τη μιζέρια και τη φτώχεια ή η εύνομη διαχείριση. Μεταξύ των δύο τι κρίνεται. Δεν πρέπει να χάνουμε όμως τις προπτικές ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μόνο βάσει των αριθμών δεν συμμετέχει ε, δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων αυτών. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρία σημεία εν ώψη αυτών των προκλήσεων. Ένα, την πυκνότητα αυτών των προγραμμάτων, δεύτερο απλούστευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και διαδικασιών χρηματοδότησης, αυτή είναι μια παλιά συζήτηση, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς ε, θεσπίζουμε προγράμματα, αλλά όταν πάμε επί τόπου να βρούμε τους ε, δικαιούχους, ε, πάντοτε υφίστανται αυτές οι ανησυχίες. Πρέπει να βρούμε μηχανισμούς που διασφαλίζουν αφενός την ομιμότητα αλλά και το δίκαιο των ετοιμάτων. Τρίτον, η μεταρρύθμιση της διαχείρισης, της καταμερισμένης διαχείρισης, όταν βλέπουμε εμεί όταν εξετάζουμε τις δαπάνες στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διότι πολλές φορές χρηματοδοτούνται μικρά σχέδια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και δεν μπορούμε εμεί σε όλα μας τα ψηφίσματα να λέμε ναι θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και της ΜΜΕ και όταν πάμε να θεσπίσουμε τους λογιστικούς κανόνες λέμε όχι, όχι είναι πάρα πολύ μπερδεμένη υπόθεση να συνεργαζόμαστε με τις ΜΜΕ ή με μικρές μονάδες. Πρέπει λοιπόν εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον νέο προγραμματισμό για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη διάρθρωση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να σας πω ε, κάτι και για την αξιολόγηση της δαπάνης. Αυτό εξαρτάται πάντα από τους ε, στόχους που ορίζουμε. Άμα δούμε τη στρατηγική 2020 για την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα, επί των πέντε στόχων μόνο δύο αφορούν το θέμα διότι το ποσοστό των απασχολουμένων μεταξύ 20 και 64 ετών ε, αντιπροσωπεύει σήμερα το 20% ενώ μια μεγάλη ενώ πολλά εκατομμύρια είναι άνεργοι. Οπότε τα δύο σημεία που τους αφορούν είναι η καταπολέμηση της στόχης, είναι η αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Χρειάζονται αυτά τα δύο μέτρα και την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Και εδώ δεν είναι ένα πρόβλημα ελέγχου προϋπολογισμού, είναι ένα θέμα πολιτικής. Και συγχωρήστε με, αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε τη στρατηγική, δεν μπο... που θέλουν τη στρατηγική τη δική μας, δεν μπορούμε εμείς να ε- εφαρμόσουμε τη στρατηγική του κυρίου Κάμερον. Στο παρελθόν το ελεγκτικό συνέδριο κατήγγειλε ότι υπήρχε μία δια... Ε, κατασπατάληση των κονδυλίων για να αξιολογήσουν και... και δεν μπορούσε να γίνει σωστή αξιολόγηση των προγραμμάτων. Εγώ θεωρώ ότι η καλή χρηματοδότηση δεν αρκεί μόνο. Χρειάζεται και η σωστή πλαισίωση, συνοχή και συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών και των των αποτελεσμάτων στους πολίτες. Σημαντικά είναι όλα όσα ε, μας δέσμευσαν για το εξάμεινο, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω στο εξής, για να είναι ωφέλιμη η κοινοτική δαπάνη θα πρέπει να έχει ένα ρόλο μουχλού. Πρέπει κατά συνέπεια να βασίζεται και στις δαπάνες που θα δεσμεύσουν τα κράτη-μέλη. Εγώ έψαξα να δω πώς τα κράτη-μέλη χρηματοδότησαν την εκπαίδευση στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας για την Ευρώπη της γνώσης. Και στον προπολογισμό της Ένωσης όμως δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος του μοχλού. Εγώ ψάχνοντας ψαχνίζοντας τον κοινοτικό προϋπολογισμό είδα ότι τα κονδύλια για την εκπαίδευση τα βρίσκουμε μόνο στον ΩΣΑ, έχουμε ναι τον έρασμο κλπ. Αλλά δεν έχουμε αυτά τα κονδύλια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχρό στις δαπάνες των κρατών μελών. Για το θέμα της κοντισιοναλίτε. Πρέπει να σας πω ότι για να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία ως ποινή για την ασέβεια των κρατών στο σύμφωνο σταθερότητας, το θεωρώ καταχρηστικότατο, διότι τελικά οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να πληρώσουν τις παρεκκλήσεις των κρατών μελών και αντιβαίνει πλήρως την αντίληψη της αλληλεγγύης που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως, το πώς τα κράτη-μέλη, το πώς Τώρα, το πώς οι περιφέρειες χρησιμοποιούν τα κονδύλια των, διαρθρωτικών ταμείων για την εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Και εκεί πρέπει να παίξει ρόλο η κοντισιοναλιτέ. Κάθε περιφέρεια μπορεί να ορίζει τη δική της στρατηγική χωρίς όμως να συμβάλλει στην Ευρώπη 2020. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο πλούσια για να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ε, επίσης διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και επί αυτού θέλω να πω επίσης μερικά πράγματα για το πώς διατίθενται αυτά τα ποσά δόθηκαν κονδύλια στην Τσεχία για την Unilever. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει στρατηγικές ε, μετατόπισης ε, των πολιεθνικών. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί εύνομη διαχείριση κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει. Τρεις παρατηρήσεις. για το θέμα της δήλωσης, το, της δήλωσης ασφάλισης. Αυτό ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία και σε άλλες χώρες. Οι συνομιλίες που είχα μου είπαν, οι συνομιλητές μου, όταν κουβεντιάσαμε για το θέμα, μου είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξαλάφρωνε ιδιαίτερα τις διαδικασίες. Και γι' αυτό που είπε η Ιούτα Χάουκ για την δυνατότητα διαχείρισης για την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεχάγης. Κάνουμε πολλά, αλλά μετά τα αγνοούμε. Η δυνατότητα ελέγχου της δαπάνης ή συλλογής ε, των φόρων. Είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά τα οποία δεν αντιμετωπίζονται σε μια ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στα κράτη-μέλη αυτό παραμένει ένα πρόβλημα. Αυτό το θέμα δηλαδή της διοικητικής ικανότητας πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και θα πρότεινα στο μελλοντικό κοινωνικό ταμείο να υπάρχει και ένα κονδύλιο για την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή διότι είτε έχουμε τότε διαφθορά ή είτε έχουμε έλλειψη δυνατότητας απορρόφησης των κονδυλίων. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα ότι εκεί όπου το ευρωπαϊκό χρήμα δεν χρησιμοποιείται σωστά και το κοινωνικό ταμείο δεν χρησιμοποιείται από το κράτος μέλος, το χρήμα αυτό θα πρέπει να ξαναδιοχετεύεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να χρησιμοποιείται για σωστά έργα, δηλαδή εφαρμογή του I want my money back. Τώρα η Φραντσίσκα Μπαλτζάνη, η συγγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2012. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά στενά το θέμα του ελέγχου και της ποιότητας της δημόσιας δαπάνης. Εγώ προσπάθησα αυτή την οπτική να την εισάγω στον προπολογισμό του 2012 και να το συνδυάσω και με τη στρατηγική διάσταση της δημόσιας δαπάνης. Θεωρώ ότι εδώ πρόκειται καθαρά για ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, για ευρωπαϊκή governance. δεν είναι μόνο το θέμα της παρακολούθησης του πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει και το σκέλος του σχεδιασμού και εκεί χρειάζεται η απόλυτη συνέργεια μεταξύ κρατών μελών και ένωσης. Οι εθνικές πολιτικές δεν σχεδιάζονται με στόχο τα κοινά σχέδια Λογικά θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα, κοινοτικά κονδύλια. Χρειάζεται κοινότητα στόχων στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και αυτό αποτελεί και την λιδία λίθο για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να προωθείται όλο ένα και περισσότερο στον κοινοτικό προϋπολογισμό και οι διαχειριστές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πρέπει να παλεύουν στην δημιουργία κοινών στόχων διότι μόνο μέσα από κοινού στόχους μπορούμε να καταλήξουμε στο κοινό, στην εκπλήρωση των στόχων του κοινού συμφέροντος, μέσα δηλαδή από την εκτέλεση κοινοτικών πολιτικών. Είπαμε κοινότητα στόχων, να σμπρώξουμε τα κράτη προς κοινού στόχους. η νομιμότητα της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων έγκυται στο ότι αυτά τα κονδύλια πρέπει να αποτελούν μοχλό που θα σμπρώχνει τις εθνικές επενδύσεις για την ολοκλήρωση κοινών πολιτικών στην επικράτεια. Με αυτήν την προϋπόθεση θα μπορούσαμε να έχουμε και αποτελεσματικούς ελέγχους. Και ο έλεγχος τι πρέπει να διαπιστώνει. Να διαπιστώνει ότι η δαπάνη εκτελείται σωστά. Ότι πληρεί το στόχο δηλαδή το κοινό συμφέρον που αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν εμείς πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σύστημα governance, ένα σύστημα διακυβέρνησης, κάθε ευρωπαϊκό εξάμεινο, που θα οθεί τα κράτη στην ανάληψη εθνικών πολιτικών που θα συμπίπτουν με κοινούς στόχους, τότε δημιουργούμε και την βάση του σωστού ελέγχου για την έπνομη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Πέρα από τους επίσημους ελέγχους που είναι δύσκολοι και που δημιουργούν πολλές φορές και έναν αντιθετικό μηχανισμό για την επαλήθευση της χρήσης του κονδυλίου. Διότι αυτό το οποίο στα χαρτιά μπορεί να φαίνεται ότι έχει δαπανηθεί με τον καλύτερο τρόπο και με τον ορθότερο τρόπο, στην ουσία μπορεί να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να μην πληρεί τον βασικό στόχο της δημόσιας δαπάνης που είναι το κοινό συμφέρον. Επίσης έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τα εθνικά κράτη και η κάθε χώρα οργανώνεται διαφορετικά στην επικράτεια όπου εμπλέκονται πολλές φορές και οι ιδιώτες και οι ιδιωτικοί μηχανισμοί στον έλεγχο της χρήσης του κοινοτικού χρήματος. Θα πρέπει όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές να τους εμπλέκουμε και στην πρώτη φάση του σχεδιασμού αλλά και στην φάση του ελέγχου Οπότε όλα τα υποκείμενα που εμπλέκονται στη χρήση του δημοσίου χρήματος θα πρέπει να εμπλέκονται και στον έλεγχο σε όλες τις βαθμίδες. Η κυρία Ρότχαστη, η οποία είναι συντονίστρια της Επιτροπής Αλίας. Να σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και τον εισηγητή για την πρόσκληση. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να διευκολύνω να παρουσιάσω τα πράγματα από τον τομέα της Αλίας στον, στην Επιτροπή Αλληλείας αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο θέμα είναι η μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας θα μεταρρυθμιστεί, θα αναθεωρηθεί. Φυσικά μπορεί τα κέντρα βάρους δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει και να τα προδικάσει εφόσον δεν έχουμε ακόμα και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναμένουμε να υποβληθεί στις 13 Ιουλίου αυτή η πρόταση της Επιτροπής. Είμαι σίγουρη όμως ότι διακομματικά στο μέλλον θα επικεντρωνόμαστε σαφώς με τον τομέα, στον τομέα της μικρής αλληλείας. Δηλαδή η τάση είναι να προαχθούν μικρές επιχειρήσεις, μικρότερες επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν και τέτοια αιτήματα όσον αφορά την πρόθεση αυτή, πράγμα το οποίο δεν θα διευκολύνει τα πράγματα για τον έλεγχο προϋπολογισμών. Όμω πολιτικά είναι σημαντικό αυτό, διότι οι μικροί αλληλεί με την αηφορία στην αλληλεία δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης από ότι η βιομηχανική αλληλεία. Εδώ πρέπει, όπω τόσο συχνά, να καταφέρουμε να πετύχουμε το απαιτούμενο, να έχουμε ένα σύστημα ευσύνοπτο για τους αλληλεί και να αποφύγουμε υψηλά επίπεδα σφαλμάτων αν έχουμε τον στόχο ευφυών λύσεων που θέλουμε να ενταχθούν, που θα αξιολογούνται στη συνέχεια και εύκολα θα μπορούν να, οδηγήσουν στα σωστά συμπεράσματα η μεταρρύθμιση στο Ταμείο Αλίας με το δεύτερο μέσο διευκόλυνσης στον τομέα της Αλίας θα συγχωνευτεί. Από το δεύτερο αυτό μέσο χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή υλοποιούνται ελεγκτικά μέτρα έλεγχη και συλλογή δεδομένων. Πολλά απομένουν να γίνουν ακόμα, διότι η κατάσταση των αλλιευμάτων στις ε, θάλασσες και η κατάσταση για αυτά τα αλλιεύματα είναι ανεπαρκής. Πέρα από όλα αυτά, από το μέσο της ε, εταιρικής σχέσης ε, και των συμφωνιών αλληλείας με τρίτες χώρες που χρηματοδοτούνται. Ιδιαίτερα αυτές οι συναλλαγές είναι ευαίσθητα θέματα, διότι ο έλεγχος των τρίτων χωρών αυτόνομα ε, γίνεται και έτσι δύσκολα μπορούμε να έχουμε μια, μια ευσύνοπτη κατάσταση. Εδώ πρέπει να μεριμνήσουμε οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίζονται. Αυτό πρέπει να ενταχθεί στις αλλιευτικές συμφωνίες και θα χαιρόμουν αν υπήρχε υποστήριξη στο αίτημα από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών διότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται, αυτά που χορηγούμε εμείς χρησιμοποιούνται όχι προς τους ορθούς σκοπούς. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο, αν θέλει να συμμετέχει στη συζήτηση. Όχι. Ο κύριος Μπάλτσιξ. Αγαπητοί συνάδελφοι των διαφόρων επιτροπών, δεν πρόκειται να επεκταθώ πάνω σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, διότι όσοι μίλησαν για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και τη δημιουργία ενός συστήματος, μίλησαν για τον στόχο της βελτίωσης της ποιότητας των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της χρήσης των κονδυλίων. Θα μιλήσω ως άτομο που επί 5-6 χρόνια ήταν υπεύθυνο για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής ε, και την χρήση των κονδυλίων σε μια μικρή χώρα, τη Λιθουανία. Ως προς την χρήση των κονδυλίων, ένα θέμα τέθηκε για τις συνεισφορές ορισμένων κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και τέσσερα άλλα κράτη-μέλη πληρώνουν πολύ περισσότερα, συνεισφέρουν περισσότερα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όσα λαμβάνουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα υπόλοιπα 22 κράτη-μέλη παρέχουν μερική υποστήριξη στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρόλο που μας αποκαλούν πολύ συχνά ε, φτωχές χώρες ε, ή ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να έχουμε διαφορετική εστίαση νομίζω στη συζήτησή μας, διότι συνεισφέρουμε κάπως τον προϋπολογισμό. Σχετικά με ένα άλλο θέμα, η λιγοτερο ανεπτυγμενες χωρες θα πρεπει να εχουμε διαφορετικη εστιαση Χάουγκ δικαίως έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υπάρχει κανονισμός σχετικά με την χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Επίτροπος έχει αναλάβει την ευθύνη να εκδώσει μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, στα κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολύ λίγα άτομα που γνωρίζουν καλά την αρχή ε, της, ε, των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της χρήσης των κονδυλίων. Υπάρχει έλλειψη γνώσεων. Τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την χρησιμοποίηση των κονδυλίων θέλουν να προστατεύσουν τις δουλειές τους. Δεν ενδιαφέρονται να πλουστεύσουν τους κανόνες ούτως ώστε να μην κατηγορηθούν ότι ξοδεύουν ακαταλήλως ε, τα, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην εκδιωχθούν. Τι θα γίνει σε μερικά χρόνια, θα διαβάζουμε και πάλι εκθέσεις, ο κίνδυνος φάλματος θα είναι κάπως μικρότερος και ακούμε, θα ακούμε προτάσεις για ενδεχόμενε βελτιώσεις στο μέλλον, αλλά η κατάσταση γενικά δεν θα αλλάξει. Ενώσο δεν αποδίδουμε ευθύνη σε υψηλό επίπεδο, θα έχουμε δυσκολίες με την χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Κύριε Πρόεδρε, επισκεφτήκαμε την Ιταλία προσφάτως και Πήραμε μερικές αποφάσεις χθες και θα έπρεπε να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ορισμένα συστήματα ε, διαδραστικά ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα και στα εθνικά όργανα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αλλαγή αυτών των αρχών και των κανόνων, ούτως ώστε να μετατεθεί ε, η ευθύνη στην Επιτροπή επίσης και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία αλλαγής θα είναι πολύ χρονοβόρα. Συμπέρασμά μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη ε, για την παροχή και παρουσίαση απλών αρχών και οι αρχές αυτές θα έπρεπε να εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια ε, πρότυπη, μια τυποποιημένη ε, διαδικασία για τους δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ συνάδελφος Ανδρέα, η συνάδελφος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην... Είμαι μέλος στην Επιτροπή και θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία ανέφερα εκεί. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο για το πόσο αποτελεσματικά δαπανώνται τα κονδύλια εκτός από τις συστάσεις ε, της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως αγνοείται αυτή η έκθεση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για πρόσθετη αξία γιατί δεν έχουμε μέτρο, δεν έχουμε γνώμονα για το πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα κονδύλια στο παρελθόν αν δούμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, τα σφάλματα που αναφέρονται δεν ενθαρρύνουν περαιτέρω διερεύνηση των κυριότερων τομέων πολιτικής. Εμείς ε, όλο και χαμηλότερα θέτουμε τον πύχη για την ποιότητα όταν γίνεται λόγος για από το μηδενικό επίπεδο σφάλματος να περάσουμε σε ανεκτό επίπεδο σφάλματος. Πολύ δύσκολο σε μια περίοδο κρίσης, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες για την παλαιότερη προηγούμενη χρήση κονδυλίων και κάτι τέτοιο καθιστά ανέφικτο αυτό το στόχο, αδύνατο αυτό το στόχο. Στη δική μας Επιτροπή ε, συχνά είχα ζητήσει αξιολόγηση για παράδειγμα του Ταμείου Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων Παγκοσμιοποίησης και χωρίς αναφορά στην Unilever που είναι ένα πολύ αρνητικό παράδειγμα επιχορηγήσεων πολύ πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα σε μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υπεξαίρεση κονδυλίων, η κακή τους χρήση εντοπίστηκε και τώρα τουλάχιστον σε κάποιες χώρες ξέρουμε ότι αυτά τα κονδύλια γνωρίζουμε καθοριστικά ότι δεν δαπανώνται με τον σωστό τρόπο. Γιατί να συνεχίσουμε να εγκρίνουμε χρηματοδότηση για τέτοιες εταιρείες που κλείνουν και απολύουν εργαζόμενους αν δεν έχουμε μέτρα και σταθμά γνώμονα να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Για το Ηνωμένο Βασίλειο θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για το πώς δαπανώνται εκεί τα κονδύλια. Γιατί όταν γίνεται ακόμα και λόγος για γενικές διακηρύξεις ή δηλώσεις, δηλώσεις ή διακηρύξεις κυβερνήσεων, πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα περισσότερα κονδύλια πάνε στις περιφερειακές αρχές. Οι ίδιες αρμόδιες ε, ε, περιφερειακές αρχές. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να τοποθετείται για την δαπάνη, για την δαπάνη αυτών των κονδυλίων. Και έχω παρακολουθήσει τέτοιου είδους προγράμματα και είδα πολλές ατυπίες και παρατυπίες. Και πέρα από αυτά είδα ότι οι φορείς που δίνονται αυτά τα κονδύλια δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διαχείρισή τους. Τούτων λεχθέντων. Πιστεύω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε και είδα ότι οι συνάδελφοί μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή και στην Οικονομική και στην ε, ε, Επιτροπή Αλίας ε, θέτουν το βάρος στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και ελπίζω ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος θα θέσει αυτός κέντρο βάρους στην χορήγηση απαλλαγής σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Τώρα φυσικά έχω τον πειρασμό να σχολιάσω την παρέμβαση της κυρίας Ανδρέας αλλά δεν θα το κάνω αυτό γιατί δεν έχουμε τόσο συχνά την ευκαιρία να συνερχόμαστε με τους ειδικού και να συζητούμε με τους ειδικού, με τους επαείοντες που σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές μας εργάζονται για αυτά τα θέματα με τη δαπάνη αυτών των κονδυλίων που προσπαθούμε να ελέγξουμε. Χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα για το ότι σήμερα το πρωί έχουμε την ε, εισηγήτρια από την ομάδα μας που μπορούμε να χαιρετήσουμε θα ήθελα δύο παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη αναφέρεται σε κοινό στόχο και έργο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτελέσει. Όταν πρόκειται για το θέμα της ποιότητας των δαπανών, μεγάλη πρόκληση στο μέλλον θα είναι η συνεργασία μας με τα εθνικά κοινοβούλια και με τα περιφερειακά κοινοβούλια να ενισχυθεί εκεί όπου υπάρχουν αρμοδιότητες στον δικό τους τομέα για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων αυτών των προγραμμάτων. Με αυτά τα περιφερειακά και hm, τοπικά κοινοβούλια θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και να εντείνουμε αυτή τη συνεργασία. Διότι πιστεύω ότι η συνειδητοποίηση πρέπει να αφυπνιστεί, η συνείδηση να αφυπνιστεί, ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δαπανώνται υπό δική τους αρμοδιότητα να αντιληφθούν ότι είναι χρήματα δικών τους φορολογουμένων και δικών τους φορολογουμένων και αυτό αξίζει να προσεχθεί, δημιουργεί μια πρόσθετη αξία. Πρόσθετη αξία και για τον έλεγχο των δαπανών. Διότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί επιτόπου αν ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια, αν ενισχύει, ενδυναμώνει την περιφερειακή οικονομία, αν βελτιώνει την κατάσταση σε σχέση με την ανεργία περιφερειακά, αν ενισχύει την περιφερειακή αλληλεία. Αυτό μπορεί και θέλει η Ευρωπαϊκή Ετροπή δεν μπορεί να τα ελέγχει ίδια. Ούτε εμεί μπορούμε να τα ελέγξουμε όσον αφορά την ποιότητα. Από πλευρά ποιότητα, εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις εθνικές αρχές, εθνικά κοινοβούλια και περιφερειακά κοινοβούλια. Να τα αφυπνίσουμε, να συνειδητοποιήσουν ότι εκεί έχουν αρμοδιότητα ελέγχου και η εθνική ε, δήλωση τότε μόνο θα αποκτήσει αξία η εθνική διακήρυξη για την χρήση αυτών των κονδυλίων. Γιατί και σε σχέση και με την αντιπολίτευση θα μπορέσει και αυτή να ε, εμπλακεί ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση εκεί πώς δαπανώνται αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια περιφερειακά. Αλλά όσον αφορά και τον έλεγχο αλλά και την ποιότητα τότε θα είχαμε πιστεύω ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός που θα μπορούσε να σημειωθεί. Μεγάλη πρόοδος. Το δεύτερο αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Το δεύτερο που θα είχα να πω. Κύριε Μπόστοκ, αν μια τέτοια στρατηγική επί της ουσίας θα την υποστηρίζατε εσεί και θα μπορούσατε να δώσετε κάποια ενίσχυση να ενδυναμωθεί, τότε θα, αυτό θα συνεπαγόταν τα εξή για το ελεγκτικό συνέδριο. Πρώτον, η συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ή με την Ομοσπονδιακή Γερμανία, με τα περιφερειακά ελεγκτικά συνέδρια των κρατηδίων θα έπρεπε να ενταχθεί στην Ομοσπονδιακή Γερμανία και να γίνει η προσπάθεια να υπάρξει κατεύθυνση για το output αυτής της στρατηγικής που θα έπρεπε να ενισχυθεί. Grazie, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής ΣΥΟΡ. Είμαι λοιπόν μέλος ε, της Αγίας Τριάδας ε, της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί η Αγία Τριάδα να έχει μεγάλη σημασία, αλλά όχι στα δημοσιονομικά θέματα ο εισηγητής ρητορικά μας είπε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron ε, πέρσι είπε ότι ε, θέλουμε ένα όριο για τον προϋπολογισμό 2011, αλλά νομίζω ότι υποστηρίχθηκε και από τις κυβερνήσεις ε, της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Δανίας, των κάτω χωρών, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ένα, μια εκπομπή ε, την γερμανική ε, τηλεόραση σχετικά με το κόμμα σας. Δεν ξέρω αν το κόμμα σας θα υποστηρίξει μια συνεχώς αυξανόμενη κατάσταση του προϋπολογισμού σχετικά με την ποιότητα των πληρωμών και των δαπανών. Πρέπει να εξετάσουμε και την φύση, την ίδια τη φύση του προϋπολογισμού. Όπως μας φαίνεται ότι τα κονδύλια ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κονδύλια που καθοδηγούνται, διευθύνονται από τις κυβερνήσεις. Θα υπάρχει πάντοτε επίπεδο σφαλμάτων. Υπάρχει και ικανότητα απορρόφησης. Και όσο μεγαλύτερο αυξάνεται το, την κάλυψη θα αυξήσετε και το ποσοστό των σφαλμάτων αν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στον προϋπολογισμό, υπάρχουν και δεν ε, ξοδεύονται, διότι κανείς δεν ξέρει πώς να τα ξοδέψει. Υπάρχουν προβλήματα συγχρηματοδότησης ή άλλα προβλήματα. Το 2008 2,8 δισεκατομμύρια επιστράφηκαν στα κράτη-μέλη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να τα απορροφήσει, να ξοδέψει τα κονδύλια αυτά. Γιατί λοιπόν μιλάμε για ανάγκη μεγαλύτερων προϋπολογισμών όσο περισσότερο οθούμε τα πράγματα, οδηγούμεθα σε ε, μια, σε μια, ε, μια ελεγχόμενη οικονομία κρατικά ελεγχόμενη σχετικά τι γίνεται με τις φτωχότερες ε, περιοχές, τις φτωχότερες χώρες. 1% νομίζω ότι είναι αρκετό. Επίσης, σχετικά με την Επιτροπή ΣΟΥΡ, sure, πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε την δομή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μετά το 2014. Πρέπει να προσανατολίζεται προς ε, το μέλλον και προς την ανάπτυξη αντί να αντλούμε συνέχεια κονδύλια. Η κυρία Μπερές μίλησε για τα διαρθρωτικά ταμεία ε, και την ομοιρία για την οικονομική ε, διακυβέρνηση σε σχετικά με τα θέματα τα οποία μιλάμε. Είπε ότι διαρθρωτικά ότι διαρθωτικά ε, ταμεία για ορισμένα κράτη-μέλη είναι μη αποτελεσματικά. Αυτό ήταν ήδη ένα χαρακτηριστικό στο ε, σύμφωνο σταθερότητας ε, και δεν χρησιμοποιήθηκε το χαρακτηριστικό αυτό. Δεν χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο για καλές δημοσιονομικές πολιτικές και το πρόβλημα του δημοσιονομικού της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι ότι τα κίνητρα δεν είναι στο σωστό μέρος και μετά διερωτόμαστε γιατί έχουμε τα κακά αποτελέσματα. Η κυρία Χάουκ παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Το βρίσκω καλό ότι μου δίνετε τον λόγο για άλλη μια φορά και μπορώ να παρέμβω πάλι. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες και πάλι στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού να δώσω. Δεν ανήκω εγώ σε αυτή την Αγία Τριάδα ανήκω μόνο στην Επιτροπή Προπολογισμών και στην Επιτροπή Σόρ. Δεν ανήκω όμω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και πρέπει κανεί ρητά και κατηγορηματικά να πει ότι στην Επιτροπή ΣΟΡ, που αμφίδρομα από κοινοβουλευτικέ ομάδε ή από κόμματα συζητούν πέρα από αυτά τα κομματικά όρια πόσο μεγάλο είναι, πόσο μεγάλος θα πρέπει να είναι ο όγκος του προπολογισμού μα όχι με αριθμητικά μεγέθη, αλλά όσον αφορά τις κατηγορίες. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχουμε ένα όριο. Και αυτό το όριο δεν μπορεί να επιβληθεί από κάποιο κράτος μέλος. Έχει καθοριστεί από τη συνθήκη. Και το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων είναι 1,23% για πληρωμέσα ε, όσον αφορά το ΑΕΠ αυτό είναι το ανώτατο όριο για το δημοσιονομικό μας πλαίσιο και σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κινηθούμε αν θέλουμε, αν επιθυμούμε. Αυτή τη στιγμή δεν το επιθυμούμε να το κάνουμε αυτό, να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Στον ενισχύει δημοσιονομικό κανονισμό αποφασίσαμε κάτι άλλο. Παρόλα αυτά όμως αυτό έχει καθοριστεί έτσι από πλευρά συνθήκη. Τώρα, όταν χρησιμοποιείτε το επιχείρημα και λέγεται το 2008 είχαμε τόσα δίσα, ε, τέσσερα δίσα, τα οποία δεν δαπανήθηκαν από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που ήταν στη διάθεσή του, δεν μπορεί κανεί απλά να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν λέει σε θέση να δαπανήσει αυτά τα κονδύλια, διότι γνωρίζουμε όλοι και εσεί το γνωρίζετε ότι 80% του προπολογισμού, 80% του προπολογισμού είναι διαχειριστική υπόθεση των κρατών μελών. <clears throat> Και εκεί είναι η αρμοδιότητα. Και δεν έχουμε κοινή διαχείριση, shared management, αλλά joint management. Δηλαδή τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για τη διαχείριση. Και όταν δεν αντλούνται αυτά τα κονδύλια από τα διαθροτικά ταμεία, τότε δεν είναι υποχρεωτικά η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού επίπεδου. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά όμως πιστεύω, πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια και τώρα ομιλεί αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού, για δημοσιονομικά από πλευρά μου. Εντάξει, παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι έργο όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όλων των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, είτε Επιτροπή Αλληλεία, είτε Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων, είτε Επιτροπή Απασχόληση, είτε οποιασδήποτε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι έργο του να μεριμνήσουν και να διασφαλίσουν πόσο προπολογισμό για ένα οικονομικό έτο που κατά τη διάρκεια αυτού του δημοσιονομικού έτου υλοποιείται και πάντα εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καλείται ως υπεύθυνη και να ερωτάτε τι κάνατε εσείς με αυτά τα οποία αποφασίσαμε εμείς το τελευταίο διάστημα ή αυτά τα οποία αποφασίστηκαν τον Νοέμβριο για παράδειγμα, τι γίνεται με όλα αυτά αυτό πραγματικά είναι έργο όλων των συναρμόδιων ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δεν είναι έργο που να μπορεί να κάνει μόνο η Επιτροπή Προπολογισμών, παρόλο που τυπικά είμαστε εμεί αρμόδιοι για την υλοποίηση του προπολογισμού. Και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού πράγματι πρέπει να μεριμνήσει πώ ε, δαπανώνται αυτά τα κονδύλια, αν βαίνουν καλώ οι δαπάνε ή όχι σε σχέση με τα κονδύλια που δαπανήθηκαν. Όλα αυτά είναι σαφή. Όταν έκανα λόγο πιο πριν ότι στην Επιτροπή, sure, α το πω έτσι, δεν έχουμε εισαγάγει ένα κεφάλι κεφάλαιο για ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό ή μια νέα δημοσιονομική τάξη των πραγμάτων, αυτό συσχετίζεται με το ότι δεν είναι δική μας δουλειά για να συζητήσουμε για αυτή τη δημοσιονομική τάξη πραγμάτων. Αλλά ενδιαφερόμαστε, είναι φυσικό αυτό και το είπαμε και το είναι γνωστό όταν διάβασε, διαβάσει κανείς την έκθεση του Σαλβαδόρ Γκαρίγα Πολιέδο, ξέρει κανείς και μπορεί να δει ότι πραγματικά θέλουμε να μεριμνήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και οικονομικοί στην δαπάνη και διαχείριση. Αλλά όταν γίνεται λόγος για απλούστευση των δαπανών, των κονδυλίων, της διάθεσης των κονδυλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν κάνουμε λόγο γι' αυτό πρέπει φυσικά, είναι αυτονόητο, να μεριμνήσουμε να μην έρχονται τα κράτη-μέλη μετά και όλα αυτά τα πράγματα να τα περιπλέκουν περισσότερο με δικές τους δημοσιονομικές τάξεις πραγμάτων που επιβάλλουν επιπλέον πάνω σε αυτούς επιπλέον, πέρα από αυτούς τους κανονισμούς και μετά να μην είναι σε θέση οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Τελευταίο σημείο, τελευταίο, Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί για αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τους επινόησε ή τους εφήβρε, αλλά όπως πάντα στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού οδηγήθηκαν σε αυτή, οδήγησαν σε αυτή τη ρύθμιση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Και θέλω να υπενθυμίσω κάτι για όλους τους συναδέλφους, για άλλη μια φορά. Εμείς υποστηρίζουμε με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, δεν υποστηρίζουμε καμιά μοναδική επιχείρηση, αλλά κατάρτιση, μέτρα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης <clears throat> προωθούνται ώστε να μπορέσουν οι άνεργοι να μπορέσουν να υποφεληθούν. Αυτά συγχρηματοδοτούμε. Θα μπορούσα να φανταστώ βέβαια ότι τα κράτη-μέλη μόνα τους θα μπορούσαν να υπομισθούν αυτή την υπόθεση. Αλλά υπάρχει το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει υπάρχουν κανονισμοί πώς μπορεί να αντλήσει κανείς κονδύλια από αυτό το ταμείο και γι' αυτό θα έλεγα είναι παρέκκληση να πει κανεί ε, ότι ε, είναι προσχηματικό να πει κανεί ότι υποστηρίζουμε τη Unilever με αυτό. Καθόλου δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς υποστηρίζουμε μόνο τους ανθρώπους που είναι άνεργοι να αντιμετωπίσουν την ανεργία αυτή στην οποία κατέληξαν. Και τελευταίο, ξέρω ακριβώς όπως όλοι, ακόμα και αν είμαι σοσιαλδημοκράτησα, ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον όγκο των κονδυλίων το πώς εμείς ε, υλοποιούμε τις πολιτικές μας. Κυρίως εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση και η χρήση αυτών των κονδυλίων που διατίθενται. Σε ποιο μέτρο και βαθμό ανταποκρινόμαστε στους στόχους που έχουμε θέσει και πρέπει να ε, υλοποιηθούν. Και βρίσκω σε αυτό το σημείο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμιά κατηγορία κατηγορία να αντιμετωπίσει. Δεν, έχει, δεν είναι ενόχο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόστοκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πλούσια και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα ε, δεν, ε, όχι να σχολιάσω για την ε, βρετανική, βρετανική πολιτική, άλλοι το έκαναν ναι. ούτε για την Αγία Τριάδα που είναι αλλού αρμοδιότητα. Ε, ρωτήθηκαν ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να βελτιώσουμε την συνεργασία με τα εθνικά όργανα, να έχουμε παραμέτρους για τα αποτελέσματα, το output Προσπαθούμε ήδη να κάνουμε πολλά σε συνεργασία με τα Εθνικά Γραφεία Λογιστικού Ελέγχου, τις Εθνικές Υπηρεσίες ε, με την Τσεχία και άλλες χώρες ε, στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας. Ε, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά στην πράξη όσο φαίνονται στη θεωρία και υπάρχουν διχογνωμίες, ε, υπάρχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα ως προς τον λογιστικό έλεγχο θέματα ε, χρόνου, συντονισμού σχετικά. Βεβαίως προσπαθούμε να ε, δούμε ποια είναι η απόδοση των λογιστικών ελέγχων, η αποτελεσματικότητά τους, να την αξιολογήσουμε. Η ικανότητα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας εξαρτάται από την σαφήνεια των στόχων που έχουν τεθεί αρχικά και στις ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί αντικειμενικοί στόχοι που δεν είναι καλά διευκρινισμένοι, τα πράγματα γίνονται δύσκολα και επανέρχομαι έτσι σε ένα θέμα από την γνωμοδότηση της, του ελεγκτικού συνεδρίου του 2010 ε, νομίζω ότι υπήρξαν θέματα κοινά στις παρεμβάσεις ενδιαφέροντα ε, και επέλεξα δύο ε, επιλεκτικότητα. Ορισμένοι είπαν ότι πρέπει να εστιαστούμε σε κοινέ δραστηριότητε πραγματικές όπου οι δαπάνε της ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν θα έλεγα ότι ε, πρέπει εκεί όπου στην πράξη να υπάρχει απλότητα και σαφήνεια. κυρία Χάουγκ ίσως ε, υπερεκτιμά την ικανότητα των κρατών μελών για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων. Είναι κάτι που μας ανησυχεί γι' αυτό αποδώσαμε ιδιαίτερα σημασία. Η κυρία Μπέρες μίλησε για την δυσκολία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να συμμορφώνονται προς τα περίπλοκους κοινοτικού κανόνες. Θέμα πρακτικό εκεί όπου πραγματικά γίνονται οι δραστηριότητες. Μας ε, βεβαίως ε, αυτά οι αλληλείς ε, έχουν να κάνουν πολλά πράγματα και πρέπει οι κανόνες να είναι κατανοητοί από αυτούς. Είναι θέμα κοινού νου. Υπάρχουν εδώ ενδιαφέροντα θέματα, υπάρχουν άτομα που φτάνουν από σημεία κίνησης διαφορετικά και θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινέ προτάσεις. Μία ή δύο σκέψεις. Υπάρχουν εδώ σκληρές επιλογές που απορρέουν από αυτή τη συζήτηση. Είναι εύκολο να είναι κανείς ε, υπέρ της καλής χρησιμοποίησης των κονδυλίων. Το κάνουμε, χρειάζεται καλή επιλογή. Συγκέντρωση στόχων, παραδείγματος χάρη διαπιστώνουμε μερικά εκπληκτικά παραδείγματα Έλλειψη συγκέντρωσης των στόχων. Εξήταζα και πάλι ε, την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το Intelligent Energy. 240 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερα ε, χρόνια 17 ε, δραστηριότητες με πάρα πολλούς τομείς στόχους. Δεν είναι νομίζω συγκέντρωση υψηλών προτεραιοτήτων. Είναι αν θέλετε πασπάλισμα, σοπουντράζ όπως λένε οι Γάλλοι. Ε, μεγάλη διασπορά. βεβαίω οι αποδέκτες ε, των χρημάτων παίρνουν λίγα χρήματα και μπορούν να πούν ότι λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει εδώ μια επιλογή ε, και μερικοί δυνητικοί αποδέκτες θα αποθαρρυνθούν αν συγκεντρώσετε την χρηματοδότηση και συγκεντρώσετε τους στόχους. Είναι θέμα πολιτικό, πολιτικών αρχών. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία λέμε ναι θέλουμε καλή προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή, αλλά σε ορισμένα πλαίσια. Αν ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό, τότε τα πράγματα γίνονται περίπλοκα και λεπτά. Τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία σκεφτόμαστε ως μηχανισμό για την μεταφορά πόρων από σχετικά ευήμερα κράτη-μέλη προς ο λιγότερο ευήμερα κράτη-μέλη, ας το πούμε έτσι αλλά πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν στα διαρθρωτικά ταμεία είναι η μεταφορά διαμέσου του προϋπολογισμού του κοινοτικού πόρων από, μία περιφέρεια ενός κρατούς μέλους σε άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους μέλους. Ε, τα διορθωτικά ταμεία μεταφέρουν πόρους από την νοτιοανατολική ανατολικη Αγγλία που είναι ε, πλούσια στην Σκοτία, ε, στην Ουαλία που είναι λιγότερο πλούσια και στη Βόρεια Αγγλία από τα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας στη Δυτική, ε, μεταφέρονται ε, κονδύλια από τη Δυτική Γερμανία. Βλέπουμε μεταφορές που γίνονται ανάμεσα στις περιοχές των διαφόρων χωρών μελών. Είναι αυτό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεν ξέρω. Επίσης, βλέπουμε ποιος είναι το ανεκτός ανεκτός φάλμα και εδώ υπάρχουν ορισμένα trade-offs που, ε, ποιος είναι υπεύθυνο για την χρήση των κονδυλίων, τι κίνδυνο μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μειώνουμε τους κινδύνους ε, με πιο αυστηρούς κανόνες. Είναι ερωτήσεις που απαιτούν δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι πολιτικό σώμα, είναι τεχνική ε, οργάνωση, όργανο και γι' αυτό θα σταματήσω πρωτού πω κάτι που δεν θα έπρεπε να πω ο συνάδελφο Χατζημαρκάκη που είναι και ο εισήγητή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ κύριε Μπόστοκ για αυτά που αναφέρατε. Ποιότητα ευθύ εξ αρχής μέσω απλούστευση και μέσω ελέγχων. Αναφέρατε το παράδειγμα της γεωργική πολιτικής. Ε, πετυχημένο αυτό. Σε σχέση με την επικέντρωση συμπίκνωση έργου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ώστε να υπάρχει ένα σωστό, ε, ένα σωστός μηχανισμός ελέγχου που θα βελτιώνει τα πράγματα όπου η ποιότητα των δαπανών θα είναι ανώτερη σε πολλούς τομείς σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Παρ' όλα αυτά η συνάδελφος Ρόντουστ προανέφερε ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκεί. Ναι, αυτό άκουσα, αυτό είπατε. Για την Αλία είπατε. Μαλία. Ναι, και τρίτες χώρες παρέκκληση χρήσης. Και παρόλα αυτά λοιπόν, δυνατότητα ή πιθανότητα παρέκκλησης της χρήσης εκεί πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Ευρωπαϊκή προσθέτη αξία, να παραμείνουμε στο παράδειγμα που προναφέρατε για την κατανομή των επιμερισμού από τις πλουσιότερες σε φτωχότερες περιφέρειες Ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Δίνω συνέχεια σε αυτό, γιατί ε, χαίρομαι διότι συνάδελφοι από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να συνεισφέρουν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Έχουμε πολλά ψεύδη τα οποία είναι διάσπαρτα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να καλύψουμε την διαφορά. Α, οι πιο πλούσιες περιφέρειες να βοηθήσουν τις φτωχότερες. Όμως δεν ανέκαμψαν οι φτωχότερες, δεν κάλυψαν την ε, απόσταση η δυνατότητα διαβίβασης ή μεταφοράς υπάρχει έστω και αν είναι σε χαμηλότερο επίπεδο αλλά σε τελικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει το ευκταίο αποτέλεσμα. Έχουμε επιχειρήσεις όμως από τον πυρήνα, από την καρδιά της Ευρώπης που πήραν πολλές παραγγελίες. Αν δούμε ποιος ε, δημιούργησε το αεροδρόμιο στην Αθήνα, μια, ευρωπαϊκή επιχεί... μια γερμανική επιχείρηση ήταν που αποκόμισε τεράστια κέρδη. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή η πολιτική συνοχή ε, δεν είναι εκείνη που πραγματικά εκφράζει εκφράζει αλληλεγγύη, αλλά είναι ουσιαστικά η διεύρυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς με άλλα, με μέσα και εργαλεία και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και Ας δούμε το παράδειγμα για το οποίο ανέφερα πιο πριν, για την Ελλάδα. Οι Έλληνες από κοινού με τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους δεν είναι σε θέση να αντλήσουν κονδύλια. Δεν είναι σε θέση να αντλήσουν κονδύλια. 30 χρόνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται πίσω από την Ρουμανία και τη Βουλγαρία, στην οποία θέση έχουν διολυστήσει σε σχέση με την ικανότητα να αντλούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολέθρια αυτή η αξιολόγηση, όχι μόνο για του Έλληνε, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι επί χρόνια ολόκληρα δεκαετίε δεν ήταν σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμού να βοηθηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση τα κράτη-μέλη. Αυτό σε ποιο συμπέρασμα οδηγεί, ότι παρακολουθούσαν με σταυρωμένα τα χέρια πώ διεφθαρμένοι πολιτικοί λαιλάτισαν τα ταμεία συνοχή και τα κονδύλια συνοχή. Και θέλω να πω ότι σε σχέση με την χορήγηση απαλλαγής, επειδή ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί και για τα τελευταία χρόνια να αποδείξει και να πει τι έγινε με τις διορθώσεις ε, των ε, ε, ελληματικών αυτών προγραμμάτων και σχεδίων. Δεν έχουν υποβληθεί αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να εξεταστούν αυτά τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό απουσιάζει ακόμα. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ομολόγησε, ομολόγησε ότι είναι τεράστια δυσκολία να δει τι γίνεται μέσα σε αυτό το λαβύρινθο κονδυλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν προς τη σωστή χρήση και να δει τα, ε, υποκατάστατα σχέδια και προγράμματα πώ θα έπρεπε να αξιολογηθούν. Έχει τεράστιε δυσκολίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Απαιτήσαμε όμω να το κάνει. Και αυτό εκρεμεί ακόμα και πρέπει να γίνει. Βλέπετε, όλοι κάναμε σφάλματα λοιπόν. Είναι πολύ καλή η εμπλοκή τη Utah Hawk που λέει το μπαλάκι είναι στα κράτη-μέλη. Εκείνα πρέπει, η δική του ευθύνη είναι και εκείνα πρέπει να δρουν. Αλλά όλα αυτά δεν οδηγούν στο να απουσιάζει η διαφάνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πει ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν σωστές επιδόσεις. Και έτσι έχουμε το μέσο πίεση, το μοχλό πίεση όσον αφορά τη διαφάνεια. Μπορούμε να διακόψουμε, να παγώσουμε την χορήγηση κονδυλίων και αυτό είναι ένα άλλο μέσο και αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί επιπλέον. Πρέπει να μεριμνήσουμε τώρα η αξιολόγηση όλων αυτών που προαναφέρθηκαν. Ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία, αποτελεσματικότητα, επιδόσεις, έλεγχη για τις επιδόσεις, όλα αυτά να γίνουν και προβλέπεται αυτό από πλευράς ε, της ε, συμφωνίας και έχει, θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει πώς φαντάζεται και πώς θα γίνουν τα πράγματα την έκθεση αξιολόγησης και η σημαντική εμπλοκή του ελεγκτικού συνεδρίου είναι σημαντική υπόθεση όχι μόνο να ε, χρησιμοποιείται η χρήση κονδυλίων αλλά και η επίδοση, η αποτελεσματικότητα και στην επίδοση. Υπάρχει ένα έγγραφο που μου έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολύ λόγο όμω. Είναι γενικό στου όρου του. Αναμένω και προσβλέπω να δούμε πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό τον έλεγχο επιδόσεων για κάθε δαπάνη θα τον υλοποιεί. Και αυτά που είπε η συνάδελφος Μπερές για το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας από την εμπειρία της ε, για την ε, κύρια αυτή κοινοβουλευτική επιτροπή της, της οποίας είναι πρόεδρος γνωρίζει τα πράγματα και έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πάρει από ένα γυμνό άντρα κάτι από την τσέπη του αφού δεν έχει λεφτά. Και για τα ταμεία συνοχή ή τα, ταμεία, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τελείω τη σκέψη για πειθαρχία. Πρέπει ευθύ εξ αρχή να καταστήσουμε σαφέ ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα σε όλα όσα κάνουν και όχι πάντα όπως το παρελθόν το έκαναν να ρίχνουν την ευθύνη σε εμά, να μεταθέτουν την ευθύνη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πειθαρχία ευθύ εξ αρχή απαιτείται, γιατί διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η ποιότητα. Και όπω είπε ο κύριος Μπόστοκ, ευθύ εξ αρχή πρέπει να διασφαλίζεται αυτό το στοιχείο. Η πειθαρχία ή ο πολιτισμό, η προσέγγιση με νοοτροπία πειθαρχημένη απουσίαζε και απουσίαζε από τα κράτη-μέλη. Συνάδελφος Μπαλτσάνη αναφέρθηκε στο κοινό συμφέρον και νομίζω πολλές φορές είναι ελληματική η κατάσταση όσον αφορά το κοινό συμφέρον. Παράδειγμα Unilever. Αλλά να πω ότι πάντα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτές οι δαπάνε θα πρέπει να αντανακλούν ένα κοινό συμφέρον. Πρέπει να είναι κάτι που συνεισφέρει προς την διασφάλιση του κοινού συμφέροντος. Πολλές φορές ε, το παραβλέπουμε αυτό, το αμελούμε αυτό. Αναφέρθηκε επίσης ε, τι γίνεται με την τοπική διαχείριση. Ευθύ εξ αρχή θεωρούσα ότι πρέπει να υπάρχει όριο σε σχέση με, το ανώτατο όριο του προπολογισμού. Πρέπει να, αποδείχνουμε, να αποδεικνύουμε ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να δαπανηθούν με καλύτερο τρόπο. Είμαι ευθυγραμμισμένο με τι παρατηρήσει σα. Συμφωνώ με αυτέ. Παρ' όλα αυτά όμω πιστεύω ότι πολλά μέσα, πολλά μέσα στην πολιτική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα από τα εθνικά μέσα. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει πραγματικά να αποδεικνύουμε ότι η ποιότητα είναι καλύτερη επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο ποιότητα. Και στι διαπραγματεύσει που από κοινού θα γίνουν, προ αυτό πρέπει να μα κινήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου συμμετείχαν. Το βρήκα πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα. Να συναντηθούμε και να συζητήσουμε για την ποιότητα όλοι μας εδώ. Θα ήθελα και πάλι να πω ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή συνεργασία και για την ρήξη των μέχρι σήμερα παραδόσεων για να είναι πάντα διπλωματική και να αποφεύγει να ονοματίσει κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό να μην είναι κανείς τόσο διπλωμάτης, να κατονομάζει τα πράγματα για να βελτιώνεται η ποιότητα. Ευχαριστώ. Μαρκάκης. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Χατζημαρκάκη. Πριν ολοκληρώνουμε με το πρώτο τμήμα, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Χωρίς να, μην επαναλάβω τα ήδη λεχθέντα, αυτή η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι όλο ένα και περισσότερο στο μέλλον θα παιχτεί η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην χρήση, αξιολόγηση και στον έλεγχο της δαπάνης των κοινοτικών κονδυλίων. Από τις έρευνες που έχουν γίνει τελευταία διαπιστώνεται ότι στην καρδιά των Ευρωπαίων πολιτών το σημείο κλειδί είναι η διαφθορά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην περιορίζουμε το τμήμα των ελέγχων είτε πρόκειται για την Κομισιόν, της Όλαφ ή του Κοινοβουλίου ή των κρατών μελών, να μην περιορίζουμε αυτούς τους ελέγχους στον επίσημό τους χαρακτήρα αυτοί οι οποίοι πράττουν την απάτη ε, είναι κυρίως οι... Ε, είναι, είναι κυρίως υπάλληλοι, είναι κυρίως η, η, η... che non è stato detto oggi ma ovviamente implicito οι καλαμαράδες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τι δαπάνε και άρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώ παίζουν οι κανόνε. Και αυτό που έλεγε ο κύριο Χατζημαρκάκη και η κυρία Μπερές, μην ξεχνάμε την τελευταία αντιπροσωπεία που είχαμε στην Ιταλία, όπου εκεί μας ανέφερε και ο εισαγγελέας ο διαπιστευμένος κατά της μαφίας μας ανέφερε το πώς η μαφία είναι αυτή η οποία προσπαθεί να βάλει χέρι στις ε, κοινοτικές ε, χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί και η εικόνα της ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έναντι των κρατών μελών. Η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως έναντι των κρατών εκείνων που παρουσιάζουν ε, σοβαρά λάθη και πολλές φορές και σοβαρές απάτες έναντι των κοινοτικών κονδύλιων. Και εντάξει η ποινή, η διακοπή της ε, χρηματοδότησης, αλλά από την άλλη μεριά, όπως είπε και μία συνάδελφος, το γεγονός ότι λόγω αμέλειας ή ικανότητες ή για άλλο λόγο δεν, το κράτος μέλος δεν χρησιμοποιεί τα κονδύλια, αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να επανέρχονται στο κοινοτικό προϋπολογισμό και να αξιοποιούνται ε, υπέρ αυτών οι οποίοι έχουν επιδείξει έναν σωστό τρόπο χρήσης αυτών των κονδυλίων. Επίσης, ε, για την Όλαφ είναι πολύ σημαντικό να καταβάλουμε προσπάθειες ούτως ώστε να γίνεται ολοένα και πιο στενή η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και κομισιών και κοινοβουλίου. Πριν ε, σας ευχαριστήσω τον κύριο Μπόστοκ του Ελεκτικού Συμβουλίου, της ε, συναδέλφους πριν λοιπόν ευχαριστήσω όλους αυτούς, δίνω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να εκφωνήσω κάποιο ε, λόγο. Ε, κυρία Κάτκο, ένα πράγμα ήθελα να επισημάνω. Ο έλεγχος ε, των δαπανών είναι έργο που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> δόθηκε με βάση τη συνθήκη. Αυτό που κάνει η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού είναι κάτι που καθορίζεται από τη συνθήκη. Όταν προσπαθεί η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού να κάνει αυτή τη δουλειά της, τότε αρνητικά το βλέπουν αυτό και εκείνοι που υφίστανται τους ελέγχους και άλλοι σε σχέση με το σώμα που ασχολούνται, ότι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εμά τους ίδιους και τις ίδιες ότι μόνο τότε πετυχαίνουμε βελτιώσεις όταν παίρνουμε αυτό το έργο στα σοβαρά. Και όταν το παίρνουμε στα σοβαρά και διατυπώνουμε τροπολογίε και βλέπουμε ότι υπάρχουν τροπολογίε που λέει, λένε για το διαθροτικό ταμείο σε σχέση με τι ε, διαπιστώσει ότι 95% των περισσότερων παρατυπιών αναφέρονται σε τρία κράτη-μέλη, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Αυτό δεν είναι μυστικό λοιπόν πια. Και τότε σε αυτό το σώμα γίνεται κάθε προσπάθεια να διαγραφεί μια τέτοια διαπίστωση. Και σε σχέση με αυτή τη συζήτηση στην οποία συμμετείχα, αυτό το έργο της καλύτερης χρήσης και δαπάνης ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά. Και είναι ωραίο και σοβαρό, αλλά πρέπει να έχουμε το θάρρος σε σχέση με τα κράτη αυτά, τους εμπλεκόμενους με τα όσα διαπιστώνουμε, να κατονομάζουμε και να ζητούμε να συναθούν ευθύνε και να υπάρχει λογοδότηση. Για διαφορετικά αν δεν γίνει αυτό θα είναι υποκριτικό αυτό το εγχείρημα, θα είναι μια υποκρισία. Πρέπει λοιπόν σαν σοβαρά να το πάρουμε για να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εντολή για τον τριημερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 και η συγγητής είναι ο συνάδελφος Χατζή Μαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η κυρία Μπαλτσάνη θα μείνει μαζί μας, διότι πρόκειται για τη δική της έκθεση επίσης και έχουμε πολύ περιορισμένο χώρο για την γνωμοδότησή μας σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 για μένα ήταν σημαντικό να τονίσω στην γνωμοδότηση αυτή ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε στόχους με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όπως είπαμε και όχι μηχανισμό για την ανακατανομή πόρων μεταξύ των κρατών μέλων. Είναι συνέχεια λοιπόν τη συζήτηση που είχαμε. Θα έπρεπε επίσης να τονίσουμε την σημασία σαφούς λογοδοσίας για τα κοινοτικά κονδύλια για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε σχετικά με την ποιότητα των δαπανών μας. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την συμμόρφωση αλλά για το βαθμό που επιτυγχάνονται τα ε, επιδιωκόμενα ε, αποτελέσματα. Είναι το θέμα της αξιολόγησης, της έκθεσης αξιολόγησης που θα πρέπει να έχουμε από το 2012. Μιλήσαμε για απλούστευση που είναι μέρος αυτής της γνωμοδότησης των δομών, των συστημάτων. Δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα βεβαίως των συστημάτων ελέγχου. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τον ρόλο της δήλωσης αξιοπιστίας που θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για ποσοστά σφαλμάτων στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί ε, σε σχέση με τα όσα είπε ο συνάδελφος Κέσλερ ότι θα έπρεπε να μην έχουμε πια διπλωματία αλλά ε, να κατονομάζουμε και να ντροπιάζουμε ανοιχτά και ε, θα πρέπει να αξιολογούμε την ε, αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των κρατών μελών. Αυτό νομίζω μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Τώρα έχουμε στα χέρια μας Έχουμε μια, ένα έγγραφο της Κομισιόν, το scoreboard, τον πίνακα βαθμολόγησης όπου η αποτελεσματικότητα κάθε κράτους μέλους αξιολογείται και έχουμε ε, μια ανακεφαλαιωτική έκθεση που θα πρέπει να αξιολογεί τα δυνατά και αδύνατα σημεία των κρατών μελών ε, στην διαχείριση και στον έλεγχό τους. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές σε συστήματα ελέγχου και θα θέλαμε να ξέρουμε τι πιστεύει η Κομισιόν σχετικά με την ποιότητα. Επίσης, και αυτό ήταν στις παρατηρήσεις του Hans Γκάιας, πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο εθνικά όργανα, εθνικές οντότητες. Έχουμε εθνικά ελεγκτικά συνέδρια τα οποία θα μπορούν να είναι ε, διαπιστευμένα σώματα, διαπιστευμένα βεβαίως από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή η ιδέα ανακύπτει κάθε χρόνο και θα ήθελα να καλέσω το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το μοντέλο που ανέφερε ο κύριος Μπόστοκ, το μοντέλο το Ολλανδικό, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Τσεχικού και να συνεχιστεί αυτή η εργασία. Επιπλέον, ε, ε, εισήγαγα δύο νέα σημεία και αυτό μπορεί να ενδιαφέρει την κυρία Μπαλτσάνη. Εάν η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει τα δημοσιονομικά, τα χρηματοδοτικά μέσα, όσον αφορά την πολιτική συνοχής πρώτα απ' όλα. Σχετικά με την πολιτική συνοχής μιλούμε κυρίως για επιδοτήσεις, για ε, επιχορηγήσεις και ξεχνούμε ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα χρησιμοποιώντας δάνεια. Έχουμε ένα όργανο ευρωπαϊκό για την παροχή αυτών των δανείων, την χορήγηση δανείων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μείγμα, μείγμα επιδοτήσεων και δανείων. Ίσως επίσης τα ομόλογα, ομόλογα έργων, τα project bonds που συζητούνται τώρα σε πολλές επιτροπές. Δεύτερον, σχετικά με την κοινοτομία και ορισμένα προγράμματα ερευνών και μας είπε ο κ. Μπόστοκ ότι ότι το πρόγραμμα καινοτομίας ανταγωνιστικότητα το πρόγραμμα Intelligent Energy που ανέφερε, εξυπνή ενέργεια, έχει ορισμένες ελλείψει. Θα μπορούσαμε ε, να βραβεύουμε καινοτομίες τεχνολογικές. Ε, έχετε ένα upfront financing για την ώρα και μετά πρέπει να αιτιολογήσετε γιατί χρειάζεστε αυτήν την χρηματοδότηση. Αλλά θα μπορούμε να σκεφτούμε να βραβεύσουμε, να επιβραβεύσουμε κάποιον που έχει μια καινοτομία. Είναι ένα μοντέλο που ε, στο Ισραήλ, ε, στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένε Πολιτείε λειτουργεί καλά, θα μπορούσε ε, να μειώσει το κόστος λογιστικού ελέγχου και τις επιπλοκές. Εφόσον δεν είχα πολύ χώρο για την γνωμοδότηση, έχω τις ακόλουθες τροπολογίες, θα εξετάσουμε την δυνατότητα βραχυτέρων ε, περιόδων προγραμματισμού, η προγραμματισμού 7 ετών καθιστά δύσκολο για μας να αξιολογήσουμε όχι μόνο την νομιμότητα και κανονικότητα, αλλά επίσης και την αποτελεσματικότητα και θα έπρεπε ε, να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει φιλόδοξες προτάσεις ούτως ώστε να υπάρχουν αυτόνομες χρηματοδοτικές δυνατότητες. Ο κύριος Λιμπαντόφσκι έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ε, Βεβαίω πολλοί δεν ικανοποιούνται στα κράτη-μέλη ε, σχετικά με αυτόν τον πρόσθετο φόρο αλλά υπάρχουν και άλλες ιδέες ίσως ε, που η Επιτροπή θα μπορούσε να λάβει υπόψη και τέλος η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα ε, να αποχαρακτηρίζει τα ε, συστήματα, τα πιστοτικά, τα εθνικά, αν δεν έχουν καλή απόδοση, αυτές οι κυρώσεις μπορεί να είναι ε, πολύ πιο αποτελεσματικές ε, από τα συστήματα που έχουμε. Εφόσον δεν είχα αρκετό χώρο, ε, έπρεπε να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τώρα ήμουνα πάρα πολύ διακριτικός. Δεν ήθελα να επέμβω σε μία συζήτηση που ξεπερνάει τα όρια μιας Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Αναφέρθηκε ο εισηγητής ε, στα πιο καυτά σημεία της, ε, των δηλώσεων του κυρίου Σεμέτα. Σίγουρα εμεί θα εργαστούμε για αυτά τα σημεία. Δεν θα αναφέρω τίποτα όμως ε, σχετικά με την απλούστευση, διότι η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα σε αυτό. Εμείς θέλουμε μία πιο ρεαλιστική λύση. Εργαζόμαστε προς στιγμή στην ε, σύνταξη των ε, τομεακών ε, βασικών πράξεων, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε απλούστερα μέσα, το output, απλούστερα μέσα που δεν θα είναι τόσο ε, εύκολα στη διάθεση ε, της ε, απάτης ή των πεθοδηγού στη δημιουργία λαθών. Όλα αυτά είναι βέβαια πολύ εύκολα κανείς να τα λέει, αλλά δύσκολα μπορεί να τα ερμηνεύει σε συγκεκριμένες πράξεις. Επί αυτού λοιπόν εργάζεται η Κομισιόν και θα ήθελ, και σας το λέω εδώ πληροφοριακά για να μην σας διαμορφωθεί η εντύπωση ότι η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα προς στιγμήν. Το λεκτικό συνέδριο θέλει το λόγο, όχι. Συνάδελφος Γκέγερ. Ναι. Ούτε από το δικαστήριο μου, ούτε από το ελεγκτικό συνέδριο. Εκείνο που θέλω είναι αυτό το σημείο υπό το 3 που ο Γιώργος Χατζημαρκάκης το ρωμαϊκό 1-3. Δεν έχω τίποτα κατά της ιδέας που βρίσκεται πίσω από αυτό συζητούμε ότι στις διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου και στις διαφορετικές ομάδες και στα ψηφίσματα όταν θέλουμε να δούμε ποια συνεισφορά είναι η σωστή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά θα επιθυμούσα σε αυτό το σημείο να βρίσκαμε μια διατύπωση που θα διευκόλυνε την αποφυγή μιας παρανόησης που φοβούμε ότι μπορεί να επισυμβεί. Δηλαδή το ότι εμείς ως ελεγκτές των προϋπολογισμών θα το χαιρετίζαμε από την άμεση επιχορήγηση στην πολιτική συνοχή να περνούσαμε σε μια άλλη ιδέα, δηλαδή σε δάνεια και πιστώσεις. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό εννοείς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε από κοινού μια διατύπωση που θα ανταποκρίνεται σε αυτό το θέμα καλύτερα. Είμαι σίγουρα, πιστεύω, ότι μέσω δανείων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσαμε πρόσθετα να δημιουργήσουμε ένα μέσο αλλά να σκεφτούμε ως ε, επιφύλαξη ότι παντού εκεί όπως για παράδειγμα στη Γερμανία όπου δημόσιες θέσεις δαπανούν κονδύλια από τα διαρθωτικά ταμεία δημόσιες αρχές και, παρο... και συναφή πιστώσεις και δάνεια λόγω της οικονομικής κρίσης του δημοσίου δεν μπορούν να αντληθούν διότι απαγορεύει την σύναψη νέων δανείων και πιστώσεων η ελεγκτική αρχή στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα λοιπόν αυτό το μέσο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν αξίζει. Και γι' αυτό για τη διατύπωση που επέλεξες έχω κάποιες επιφυλάξεις Γιώργο Χατζημαρκάκη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι προσκαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο να χρησιμοποιεί αυτό το μέσο. Όχι. Είναι ένα συμπληρωματικό μέσο, μάλιστα, αλλά προ όφελο τη πολιτική συνοχή. Και μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό το στόχο. Αν έχουν πολύ λίγο καλύψει τι διαφορέ οι περιφέρειες όπω πιο πριν ανέφερε στην τοποθέτησή σου αλλά το μέσο των πιστώσεων και δανείων στην πολιτική συνοχής να το διατηρήσουμε, αλλά σε σχέση με την εντολή που θα δινόταν να μην προχωρήσουμε μέχρι εκεί. Θα έπρεπε περισσότερο να γίνεται χρήση ενός τέτοιου μέσου συμπληρωματικά. Γι' αυτό η διατύπωση είναι σημαντική υπόθεση εδώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφος Χατζημαρκάκης. Για το θέμα ή την επισήμανση αυτή είμαι ευγνώμων, διότι δίνει ευκαιρία να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται από τα πλεονάσματα που υπάρχουν να χρησιμοποιηθεί η μόχλευση Hebel effect, leverage, leverage, μοχλευτική επίπτωση, δηλαδή όσον αφορά την risk shared facility, δηλαδή τον επιμερισμό κινδύνων σε σχέση με αυτό το μέσο. Εκεί ένα δις από το πρόγραμμα για την έρευνα ε, που διατίθεται και από αυτό καταλήγουμε με την μόχλευση μέσω της ε, ε, ιδιωτικής αγοράς κεφαλαίων που μπορούν να, μπορεί να οδηγήσει στην άντληση περαιτέρω δυνατοτήτων και μπορεί έτσι να απαμβληθεί ο κίνδυνος. Αυτό θέλουμε ακριβώς να γίνεται ως, επίπε, ως ε, μοχλευτική επίπτωση στον τομέα της συνοχής. Είμαι ευγνώμων για την επισήμανσή σου. Να βρούμε τη σωστή διατύπωση ώστε αυτό το επίπεδο μόχλευσης να επιτευχθεί σωστά. Ευχαριστώ. Grazie. Volevo ricordare che per να σας θυμίσω ότι 18 Απριλίου 2011 στις 12 η προθεσμία για τις τροπολογίες. Πάμε στο σημείο 17, ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, εισηγητής ο συνάδελφος Καοπίν, ο οποίος μας είπε ότι μπορεί να δεχτεί μόνο στις 11. Θα κάνουμε λοιπόν ένα τέταρτο διάλειμμα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι

Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. ζητώ να καθίσετε. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τον ε, εισηγητή μας και φτάνουμε ε, στο σημείο 17 ε, της ημερήσιας διάταξης δίνω στον λόγο στον εισηγητή Ιβάιλο Κάλφιν και καλωσορίζω τον κύριο Ντεβρή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να με συγχωρήσουν όλοι οι συνάδελφοι που περίμεναν για μένα. Νόμιζα ότι το σημείο αυτό θα φτάσει πιο αργά στην, στο πρόγραμμά σας. Λυπούμε που σας άφησα να περιμένετε. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας εργάζεται αποτελεσματικά. Αυτή η έκθεση η οποία ε, προετοιμάστηκε εδώ και μερικό χρόνο που εστιάζεται στις ε, δαπάνες για ε, το νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης σε τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Γεωργία. Η ιδέα της έκθεσης ήταν μέχρι ποιου σημείου τα κονδύλια έχουν δαπανηθεί αποτελεσματικά, πώς σχεδιάστηκαν τα προγράμματα, ε, ποια ήταν η υλοποίηση ε, στον πρώτο χρόνο που οδήγησε σε επιτεύγματα επιτυχημένα και πώς αξιοποιήθηκαν τα μέσα βάσει των, ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Η έκθεση και θα ήθελα να συγχαρώ το ελεγκτικό συνέδριο ε, για αυτό το, την έκθεση ε, διότι έχει διάφορες ε, επιθυμίες που θα λάβουμε υπόψη στις μελλοντικές μας αποφάσεις για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για νέα μέσα, βεβαίως κάθε νέα πρωτοβουλία θα απαιτήσει ε, κάποιο χρόνο προσαρμογής ούτως ώστε να αποδώσει καλύτερα, αλλά ε, μπορούμε να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εν τω μεταξύ, μετά την ε, προετοιμασία της έκθεσης υπήρξε αλλαγή στην Επιτροπή. Έχουμε την, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά ε, είναι η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του μηχανισμού γειτονίας και εταιρική σχέση. Είναι ο Επίτροπος Φούλε που είναι η αρμόδιος και υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Ποια είναι τα προβλήματα. Είναι μικρά προγράμματα, μικρά έργα ε, με υποστήριξη δημοσιονομική και είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Ξέρω ότι έχει συζητηθεί το θέμα, αλλά ίσως έχουμε τη δυνατότητα να ε, αναθεωρήσουμε και πάλι. Ξοδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοσιονομική υποστήριξη, δίνει κονδύλια για τον προϋπολογισμό έναντι της επίτευξης ορισμένων αποτελεσμάτων και επίσης χρηματοδοτεί ε, ορισμένα προγράμματα. Νομίζω ή χρηματοδοτεί ορισμένα προγράμματα και οι δύο μέθοδοι έχουν ε, τα επιχειρήματα υπέρ. Νομίζω ότι στο Νότιο Κάφκασο τα περισσότερα κονδύλια διοχετεύτηκαν για δημοσιονομική υποστήριξη, δηλαδή κονδύλια για τον προϋπολογισμό των αποδεκτριών χωρών Βεβαίως ε, πρέπει να επιτύχουν ορισμένα αποτελέσματα, αλλά και πάλι όταν αρχίζει, άρχισε αυτή η διαδικασία, το ενδιαφέρον και η προσπάθεια ε, της Κομισιόν είναι τελικά να υλοποιηθούν τα έργα, τα προγράμματα, που, πράγμα που δημιουργεί ορισμένα προβλήματα για την επίτευξη αποτελεσμάτων από τις αποδέκτριες χώρες. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με τις προτεραιότητες που έχουν επιλογή. Πρόκειται για προτεραιότητες που εκπονήθηκαν μαζί με τις δικαιούχους χώρες, ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλούμε ότι θα υποστηρίξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν που μαζικά παράγει και εξάγει πετρέλαιο και διαθέτει πολλά αποθέματα πετρελαίου αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι θετικό και ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διερωτώ με ποιο ενδιαφέρον θα επιδείξει η χώρα για να αναπτύξει τέτοια προγράμματα και έργα. Και αυτό που διαπιστώνουμε στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν είναι ότι το πρόγραμμα αυτό προχώρησε βραδύτατα, με πάρα πολύ ε, μεγάλα κενά ανάμεσα στα διάφορα κομμάτια, στα διάφορα τμήματα, διότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Αρμπατζάν δεν είναι τόσο μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν η επιλογή κριτηρίων και προτεραιοτήτων ε, να γίνει πολύ καλύτερα. Ένα άλλο θέμα το οποίο διαπιστώθηκε στην έκθεση είναι ότι αν δίνουμε δημοσιονομική στήριξη βασιζόμαστε στις δημοσιονομικές διαδικασίες της αποδέκτριας χώρας ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια. Και εδώ έχουμε μια ανισότητα με τις ικανότητες των αποδεκτριών χωρών να συμμορφωθούν στα πρότυπα, στους κανόνες. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε πάρα πολύ τις χώρες. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Έχουμε ορισμένε ικανότητες, δικανότητες στην γραφειοκρατία, στην δίκηση, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς όταν, ότι όταν παρέχουμε δημοσιονομική ε, στήριξη σε χώρες ε, που κάνουν αλλαγές ε, στην διοίκησή τους, που επιτελούν πρόοδους για να επιτύχουν καλύτερους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν έχουμε τα ίδια πρότυπα όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η κατάσταση στις τρεις αυτές χώρες και διαπιστώνεται στην έκθεση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Και πάλι πιστεύω ότι εν κατακλείδη εστιάστηκα σε ε, μερικά από τα μειονεκτήματα του προγράμματος. Νομίζω ότι στο σύνολό του το πρόγραμμα είναι θετικό και έχει πολιτικό νόημα, αλλά ίσως θα πρέπει άλλη μια φορά να αναθεωρηθεί για να, και να ε, εξεταστεί για να δούμε τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί, ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο μεταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ένα πρόβλημα με την δημοσιονομική στήριξη είναι η ορατότητα. Κατά πόσον τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά ή έχουν άμεση σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες φορές, παραδείγματο χάρη, όταν είχαμε στην Αρμενία ανακαίνιση ορισμένων ε, κτηρίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις εθνικές προσπάθειες και τις κοινοτικές προσπάθειες ε, λόγω του γεγονότος ότι έχουμε ένα καλά επιπλωμένο κτίριο, αλλά η μόνωση δεν υπάρχει ή γίνεται με ένα παλιό σύστημα θέρμανσης. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν τα καλά αποτελέσματα και μειώνουν την ορατότητα, την γνωστοποίηση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν το μέσο αυτό του μηχανισμού που είναι πολύ καλό, πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει ίσως να ε, έχει καλύτερο συντονισμό και από ό,τι ξέρω στην ε, Επιτροπή και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καταβάλλονται προσπάθειες προς το σκοπό αυτό μετά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη στοχοθέτηση και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ε, δημοσιονομική στήριξη και την χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων και προγράμματος ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον κύριο Γκρίς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα εισαγωγικά σχόλιά του και την καλά διαρθρωμένη έκθεση και να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Φιούλε ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Είχα όμως μια συνομιλία μαζί του και επέδειξε κατανόηση για ορισμένα από τα θέματα τα οποία ανέφερε το ελεγκτικό συνέδριο και δεσμεύθηκε να τα λάβει υπόψη της παρατηρήσεις αυτής στην αναθεώρηση της πολιτικής αυτής. Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία της έκθεσής μας. Πρώτα, την περιπλοκότητα ε, της ε, πολιτικής γειτονίας και τις ανομαλίες που βλέπουμε ανάμεσα σε ορισμένα μέσα που χρησιμοποιούνται και μερικά σχόλια για πρακτικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο, η υλοποίηση της πολιτικής αυτής από την Κομισιόν στον Κάφκασο χαρακτηρίζεται από τρία επίπεδα περιπλοκότητας. Πρώτον, για κάθε χώρα εταίρο ε, δεν ε, έχουμε πέντε μέσα για την υλοποίηση της ε, πολιτικής. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας, το πρόγραμμα δράση, το στρατηγική έκθεση της χώρας, το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Επίσης, κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικό χρονικό ορίζοντα Έχουμε το πρόγραμμα δράσης μέχρι το 2011, το στρατηγική έκθεση με το 2013 και το ενδεικτικό πρόγραμμα μέχρι το 2010. Τρίτον, τα προγράμματα είναι ευθύνη διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής. Ο προγραμματισμός διαμέσου ε, του προγράμματος δράσης, του στρατηγικής έκθεσης ενδεικτικού προγράμματος είναι ευθύνη, ήταν μέχρι τώρα ευθύνη ε, της Γενικής Διεύθυνσης ΡΕΛΕΞ ενώ ε, του ετήσιου προγράμματος δράσης και τα χρηματοδοτικά ε, συμφώνια, οι συμφωνίες είναι του τομέα της Europe Aid. Αυτό έχει το τίμημά του αυτή η περιπλοκότητα. Το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε αδυναμίες μεταξύ των προγραμμάτων διότι δεν έχουμε αρκετή σαφήνεια στον προγραμματισμό και ανεπαρκείς ε, προτεραιότητες Νομίζω ότι το ενδεικτικό πρόγραμμα προσθέτει λίγα στην στρατηγική έκθεση της χώρας. Χρειάζονται ανανέωση και απλούστευση τα μέσα και οι διαδικασίες αυτές. Τη διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού χρειάζεται πολύ χρόνο, πάνω από δύο χρόνια πριν από την έγκριση του πρώτου ετήσιου ε, προγράμματος δράσης. Ο λόγος είναι οι εσωτερικές διαδικασίες ε, στις ε, δύο γενικές διευθύνσεις, RELEX και Europe Aid και αυτές οι αναβολές ε, ε, αποτελούν κίνδυνο σχετικά με την ε, συνάφεια, την χρησιμότητα της βοήθειας. Μια δεύτερη διαπίστωση είναι οι ανομαλίες μεταξύ των διαφόρων εγγράφων πολιτικής, προτεραιότητες που αναδιατυπώνονται, οι τομείς που επελέγησαν από την EuroPaid δεν προέκυψαν αρκετά σαφώς από τα προγράμματα στρατηγικής που είχε ετοιμάσει η Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ. χάρη στην Αρμενία η εκπαίδευση επελέγει από την Europaid ως βασικός τομέας, αλλά κανένα από τα τρία στρατηγικά έγγραφα που ετοίμασε η DG Relex δεν τόνισε τον τομέα αυτό. Κρύβεται μεταξύ των 25 στόχων των 7 υποπροτεραιοτήτων του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος. Στο Αζερβαϊτζάν η Γενική Διεύθυνση Europaid επέλεξε ε, την δημοσιονομική ε, βοήθεια αλλά όπως εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Αζερβαϊτζάν τόνισαν στο ελεγκτικό συνέδριο, προτιμά η χώρα την τεχνική βοήθεια. Νομίζω ότι ο, ο εισηγητής μίλησε για την δημοσιονομική υποστήριξη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα πω ότι ε, στην συζήτηση που είχατε χτες με συνάδελφό μου, και για την ε, γενική διαχείριση της δημοσιονομικής στήριξης δεν μπορώ να πω ότι τα συμπεράσματα που είχατε ε, σχετίζονται αποκλειστικά με τον Κάφκασο, αλλά υπάρχει ένα σημείο ότι η Επιτροπή δεν αποδίδει ιδιαίτερη τόση μεγάλη σημασία όταν ε, δίνει δημοσιονομική στήριξη ε, στις απάτες και στην διαφθορά. Πρέπει να είμαστε σαφείς για τους μηχανισμούς που θα πρέπει να υλοποιήσει η αποδέκτρια χώρα για να καταπολεμήσει την απάτη και την διαφθορά ε, είδαμε ότι αυτό δεν είναι πάντοτε η περίπτωση. Και κλείνω την παρένθεση. Ένα μέσο που θα μπορούσε να υποφεληθεί από την απλούστευση είναι ε, το πρόγραμμα ε, δράση. στην Γεωργία. Έχουμε 306 ειδικέ δεσμεύσεις με 64 δράσεις προτεραιότητας και 242 πρόσθετες δράσεις μπορούμε ειδικαίω να πούμε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει πάνω από 300 δεσμεύσεις ε, και ε, υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν 64 προτεραιότητες δεν είναι πολύ χρήσιμο. Ε, τρίτον, τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Το συνέδριο ε, ε, διαπίστωσε ότι είναι μεικτά τα αποτελέσματα, ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Αρμενία επηρέασε θετικά και ενίσχυσε τις μεταρρυθμίσεις. Στο Αζερβαϊτζάν δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε πρόοδος στον τομέα της ενεργειακής μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα διαχείρισης δημοσιονομική στη Γεωργία προόδευσε, αλλά όχι το πρώτο έτος, αλλά όχι το δεύτερο. Στην Απχάζια επίσης ε, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Βεβαίως, η έκθεση είναι αν θέλετε ε, μια στιγμιαία αποτύπωση του τι συμβαίνει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Πάντοτε, πάντως ε, το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να μεταρρυθμίσει την διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, απλουστεύοντας τις διαδικασίες και τα μέσα. Δεύτερον, ότι θα έπρεπε να είναι πιο επιλεκτική όταν παρέχει ε, τομεακή δημοσιονομική στήριξη. Και τελικά ε, στόχος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν πάντοτε να διαπιστώνει τα γεγονότα έτσι όπως έχουν και να κάνει πρακτικές συστάσεις. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει πλήρως επιτύχει το στόχο του, θα πιστεύω ότι η Επιτροπή θα το επισημάνει αυτό. Ε, η Κομισιόν στις απαντήσεις, στις εκθέσεις ε, του συνεδρίου θα πρέπει να περιορίζεται σε σχόλια συνοπτικά. Ε, η απάντηση των 22 σελίδων είναι ίσως υπερβολική. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεφρίς. Τέσσερις σας ζητούν να σχολιάσω για μια ολόκληρη σειρά θεμάτων και συστάσεων να ρωτήσω, θέλει να αντιδράσει και να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα όσα αναφέρθηκαν. Η Επιτροπή παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μονάρο είναι το όνομά μου. Πρώην για την Europaid όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Γειτονία και για το 2007. Θα ήθελα να σας ε, πρώτα να πω ότι εκτιμούμε και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία που είχαμε με το ελεκτικό συνέδριο σε σχέση με αυτή την έκθεση και πέρα από τις ε, τόσες σελίδες ε, σχόλια αντανακλώνται θα έλεγα υπό το πρίσμα μας ε, οι συνιστώσεις ενός θετικού εγχειρήματο και θέλουμε πραγματικά να πορευθούμε όσον αφορά αυτές τις προτάσεις και συστάσεις. Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω την σφαιρική και σωστή περίληψη που μόλις δόθηκε από τον εισήγητη θέτοντας δύο πράγματα στο επίκεντρο. Πρώτον, αναφέροντας ότι παρόλες ε, τις προκλήσεις και δυσκολίες που υπάρχουν, παρόλα αυτά αυτό το εγχείρημα ήταν θετικό. Ήταν μια θετική εμπειρία και καλό θα ήταν να πει κανείς ότι σημειώνονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όροι υπό τους οποίους ξεκινούν τέτοιες πρωτοβουλίες σε αυτές τις ε, τρεις χώρες στο Νότιο Κάφκασο. Σε όλα αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα πιο πέρα ότι πραγματικά η έκθεση με την χρησιμότητα και την σκοπιμότητά της μια περιορισμένη εικόνα δίνει στον χρόνο και στο εύρος όσον αφορά τις χώρες αυτές για το τι γίνεται σε σχέση με αυτή την γειτονία. Οδηγηθήκαμε σε 17 χώρες τα τελευταία, όχι μόνο δύο, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός στο να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα τα οποία θα διευρυνόντουσαν γενικότερα για το πώς λειτουργεί σφαιρικά η πολιτική για τη γειτονία, η πολιτική γειτονίας. Αναγνωρίζω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις όσον αφορά την δημοσιονομική συνδρομή ο εισηγητής και σίγουρα από πλευράς Επιτροπής συνειδητοποιούμε, αναγνωρίζουμε ότι με τον τρόπο που παρουσιάζεται το πολιτικό μείγμα για την δημοσιονομική συνδρομή, για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τις κυβερνήσεις και όσον αφορά και συμπληρωματικά με την πραγματογνωμοσύνη και σε σχέση με τα σχέδια και προγράμματα που καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο εύρος ε, κύριων θεμάτων είναι κάτι που θα έπρεπε να αντανακλάται στα προγράμματα και στις δράσεις αυτές. Ε, όμως σε σχέση όχι με αλλαγή του μείγματος αλλά για την επεξήγηση των σκέψεων που βρίσκονται των επιχειρημάτων που οδηγούν σε αυτό το μείγμα. Αναφερθήκατε σωστά στην πτυχή της ευδιακριτότητας, του ευδιάκριτου χαρακτήρα είναι κάτι το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά για την επιλογή της ε, πολιτικής ε, γειτονίας από τότε που ξεκίνησε έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένες προτεραιότητες και να υπάρχει συναρμοδιότητα από πλευρά των κυβερνήσεων και μια τέτοια δυνατότητα ήταν το να υπάρξει ένα εύρος προγραμμάτων μέσω των κυβερνήσεων που θα τύχανε συνδρομής Ίσως να αναφερθώ στις δύο συστάσεις που μόλις διατυπώθηκαν από τον κύριο Ντεφρίς όσον αφορά και το ελεγκτικό συνέδριο επίσης για τον προγραμματισμό. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο αναγνωρίζω βέβαια ότι το ελεγκτικό συνέδριο πολύ σκόπιμα υποβάλλει αυτές τις προτάσεις στη σωστή συγκυρία και σε σχέση και με την Ρέλεξ και την ε, υπηρεσία ε, διπλωματικής δράσης, εξωτερική υπηρεσία, διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμιστεί και ο συνάδελφος εκ δεξιών μου από την διπλωματική υπηρεσία, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, θα μπορούσε και αυτός να τοποθετηθεί. Είναι κάτι που μάλιστα αναγνωρίζουμε θετικά και θα προσπαθήσουμε στην επόμενη γενεά προγραμμάτων Ευρωπαϊκή Γειτονία να εντοπίσουμε τα διάφορα διαστρώματα για τέτοιου είδους προγράμματα και να επικεντρωθούμε πιο εξειδικευμένα στις δράσεις όσον αφορά μια συγκεκριμένη μερίσια διάταξη, μια συγκεκριμένη ατζέντα. Αλλά αυτά τα προγράμματα δράσης, αυτές οι ημερήσιες διατάξεις πρέπει να ιεραρχηθούν, να τύχουν προτεραιοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε κέντρο βάρους δράσεων και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα, συνοχή, συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων γειτονίας και των πολιτικών στόχων ώστε η οικονομική, η δημοσιονομική συνδρομή να είναι η πιο αποτελεσματική. Για το δεύτερο θέμα, για το πώς θα είμαστε πιο επιλεκτικοί όσον αφορά την ε, οικονομική σύνδρομη, με τα κονδύλια που δημοσιονομικά διαθέτουμε θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τα όσα είχαν, το, είχε τοποθετηθεί πιο πριν ο εισηγητής 50% που περνάνε μέσω του προϋπολογισμού για την ευρωπαϊκή γειτονία, αφήνοντας 30-50% περιθώριο για χρηματοδότηση για την τεχνική σύνδρομη και ε, γενικότερα προγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μείγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο και νομίζουμε ότι είναι το σωστό. Αλλά στις επιμέρους χώρες θα μπορούσαν να υπάρχουν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις και αυτό το πολιτικό μείγμα θα μπορούσε καλύτερα να επεξηγείται από πλευράς προσέγγισης και σύλληψής του και να συνδέεται με τα αποτελέσματα που προσπαθούμε να πετύχουμε με τα επιμέρους μέσα που, μας, έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα αυτά τα θέματα θα αναφέρονται σε δύο ανακοινώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει και έγινε αναφορά και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική συνδρομή, την οικονομική συνδρομή που θα καλύπτει και την γενικευμένη, την γενική οικονομική συνδρομή αλλά και την εξειδικευμένη τομεακά ε, δημοσιονομική συνδρομή. Προετοιμάζονται αυτά και θα τεθούν υποσυζήτηση κατά το δεύτερο εξάμεινο αρκετά σημεία θα αναφέρονται στις, ε, στους και προϋποθέσεις ε, που ενισχυμένα θα ισχύουν, ενισχυμένη διαφοροποίηση και το ε, κατάλληλο μείγμα με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία αυτά στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ήδη. Αν επιτρέπετε Πρόεδρε να πω τέλος ότι σε σχέση με το σχέδιο σύστασης τις συστάσεις που είδα στο έγγραφο. Φυσικά είναι δικό σας έγγραφο και δεν θέλω να αναμειχθώ στις δικές σας αρμοδιότητες όσον αφορά αυτό. Όμως πρόσεξα ότι κάποιες διατυπώσεις, δηλαδή ανησυχείτε βαθιά για τις διαδικασίες και βρίσκεται απαράδεκτο, λέει, τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε σε δημοσιονομική συνδρομή, είναι διατυπώσεις που δεν αντανακλώνται ούτε στις γενικότερες συζητήσεις που είχαμε με το ελεγκτικό συνέδριο και νομίζω πάνε αρκετά μακριά, υπερβολικά μακριά κάποιες ε, συστάσεις με, αυτή, με τέτοιες διατυπώσεις. Και σε σχέση και με την σύνοψη από πλευρά εισηγητού, νομίζω ε, και την παρουσίαση των δικών του θέσεων δεν αντανακλώνται έτσι. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσω και με αυτά τα δύο σχόλια να αναγνωρίσω την χρησιμότητα της έκθεσης και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε θετικά να αντιδράσουμε στις κύριες συστάσεις ε, που διατυπώνονται στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως κάποιος θέλει ε, να μιλήσει ε, εκ μέρους της Ρελέξ. Όχι. Τότε ανοίγω την ε, συζήτηση. Ε, η κυρία Γκρέσλερ θα ήθελε να μιλήσει νομίζω εκ Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κρίμα είναι το ότι η εξωτερική υπηρεσία, η διπλωματική υπηρεσία δεν λέει τίποτα. Διότι πραγματικά θα προσδοκούσαμε να ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτησή της. Πώς βλέπει η εξωτερική υπηρεσία, η διπλωματική υπηρεσία τα πράγματα και ποιες τροποποιήσεις, αλλαγές πρέπει να επέλθουν στο μέλλον με τα όσα μας ανέφερε ο, ο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ποια μαθήματα μπορούν να συναχθούν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό σε σχέση με τις ε, τοποθετήσεις του ε, σώματός μας. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των ενδεικτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ε, δράσης. Ποιες είναι οι απόψεις σας σε σχέση με αυτό το σημείο, αλλαγές που πρέπει να επέλθουν. Θα ήθελα να ακούσω αυτά τα στοιχεία, διότι δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα αλλάξει και με ποιο τρόπο Τέσσερα βήματα για τον προγραμματισμό θα υπάρξουν. Τα τρία βρίσκονται στην διπλωματική υπηρεσία, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το τέταρτο, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και πρέπει εκεί όταν εξειδικεύονται τα πράγματα και το, το τέταρτο, η συγκεκριμένη διαμόρφωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα γίνει. Ερωτώ και πάλι, πώς έχετε υπόψη να τα διαμορφώσετε στο μέλλον αυτά. Ποιος θα κάνει τι, ποιος θα καθορίζει τι πράγμα, ποιος θα καθορίζει ποιος θα είναι αποδέκτης αυτών των κονδυλίων. Και μετά σε σχέση με τους πρόσφυγες, αυτή ήταν η πρώτη ερώτησή μου, σε σχέση με τα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο, είχαμε μία επιστολή έξι πρέσβεων, έξι μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μια μετάθεση των κονδυλίων από την πολιτική γειτονία θέλουν να υπάρξει προ τον χώρο του Νότου, προς τη Μεσόγειο. Ποιε σκέψεις έχετε εσείς ε, και σας απασχολούν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε επιπτώσεις θα υπήρχαν από το 2014 σχετικά. ποιε επιπτώσεις ακριβώς σε σχέση με την πολιτική γειτονία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και του εισηγητή και χαίρομαι που έχουμε κάποιο χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις αδυναμίες που ακούσαμε ανεπαρκή σαφήνεια, ανεπαρκή ε, προγραμματισμός, έλλειψη συντονισμού κλπ. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό μας εκπλήσει διότι η Κομισιόν δεν είναι η πρώτη εμπειρία στον τομέα αυτό, στον τομέα της χρηματοδότησης και της υλοποίησης τέτοιας χρηματοδότησης με τρίτες χώρες. Είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς γιατί και πάλι έχουμε τα ίδια θέματα που ανακύπτουν. Θα ήθελα επίσης να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τον έλεγχο του τι συμβαίνει και του πώς ξοδεύονται τα χρήματα στις χώρες αυτές όπως ακούσαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε ορισμένες ε, περιπτώσεις υπάρχει απάτη και διαφθορά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η χρηματοδοτική στήριξη τρίτων χωρών ε, πρέπει να χρησιμεύσει για να τους μάθουμε πώς να ξοδεύουν σωστά, ορθά ε, τα χρήματα, να έχουν διαφάνεια, έλεγχο και να έχουν καλές ε, διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα, να επιμένουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Τελειώ γελιοποιούμεθα. Δίνουμε χρήματα και δεν παρακολουθούμε και δεν ενδιαφερόμαστε τι συμβαίνει με τα κονδύλια αυτά. Θα επιμένω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στην αλλαγή της μεθόδου ούτως ώστε ε, να είναι καλύτερη η χρηματοδότηση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Κανένας άλλος δεν ζητάει τον λόγο. Θα ζητήσουμε από τον εισηγητή, κ. Κάλβιν, αν θέλει να αντιδράσει, διότι ε, Είδα ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι, έχει μεγάλη ανησυχία και ότι έχει διαφορές με την Επιτροπή. Ακούθηκε ε, πάρα πολύ η λέξη διαφθορά, ε, η ανεπάρκεια σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η διατύπωση στην έκθεση έχει επιλεγεί με προσοχή και σωστά. Μιλάμε για τις αδυναμίες μέσα στην Κομισιόν. Νομίζω ότι λαμβάνονται μέτρα και αυτό ε, θα είναι σημαντικό. Δεν, ε, το Κοινοβούλιο λοιπόν ανησυχεί, ανησυχεί όταν δεν υπάρχει συντονισμός μέσα στην ίδια την Κομισιόν Ελπίζω ότι τώρα η ύπαρξη της υπηρεσίας εξωτερικής ε, δράσης θα βελτιώσει, όχι θα επιδεινώσει το συντονισμό. Υποστηρίζω τα όσα είπα ο εκπρόσωπος της Κομισιό ότι καταβάλλονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή σχετικά με τον απαράδεκτο τρόπο ε, δαπανών με τον οποίο ξοδεύονται τα κονδύλια. Αυτό αναφέρεται ε, στον προκαταρκτικό υπολογισμό ή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να ξοδεύουμε κονδύλια χωρίς να ξέρουμε ποια είναι τα αναμενόμενα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η Κομισιό θα πρέπει ενδελεχώς να αναθεωρήσει ε, να εξετάσει την χρήση των διαφόρων μέσων που είναι διαθέσιμα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ε, Γειτονίας. Λέχθηκε ότι θα μας εξηγήσει καλύτερα η Κομισιόν. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό, αν θα κρατηθεί η ίδια ισορροπία. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ε, πρόβλημα ε, με την, τις σωστές δεσμεύσεις από πλευράς των κυβερνήσεων με το twinning. Νομίζω ότι η δημοσιονομική υποστήριξη είναι πιο εύκολη από απόψε, απόψεως της γραφειοκρατικής ε, του προσωπικού, ενώ χρειάζεται πρόσθετο προσωπικό ε, για να εργαστεί στα γραφεία της ευρωπαϊκά στις χώρες αυτές για να παρακολουθεί τα προγράμματα και τα έργα, την υλοποίησή τους. Η επιλογή των μέσων θα πρέπει να βασίζεται σε μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Νομίζω ότι στις αλλαγές που προτείνει η Κομισιό αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και πάλι πρόκειται ε, για έναν έλεγχο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο που ενδελεχώς και προσεκτικά έκανε τη δουλειά του. Ε, είμαστε στις αρχές της, ε, ήταν οι αρχές της χρησιμοποίησης αυτού του μέσου. Ελπίζω να υπάρξει βελτίωση και περιμένουμε από την Κομισιό να μας δείξει ότι θα έχουμε καλά παραδείγματα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν από τα διδάγματα που θα αντλήσουμε για να μην επαναληφθούν ε, τα ίδια ασφάλματα. Ευχαριστώ τον ε, κύριο εισηγητή. Η κυρία Γκρέσλερ όμως ε, έθεσε ερωτήσεις και ίσως θα έπρεπε η Κομισιόν να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Έχουμε την ερώτηση του ποιος θα κάνει τι και δεύτερον ε, πρόσφυγες στην ε, Μεσόγειο. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τις ε, προτεραιότητες μας σε σχέση με αυτήν την κατάσταση. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να απαντήσει στις δύο αυτές ερωτήσεις. Αν συμφωνείτε να δώσετε απαντήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επανέλθουμε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Θα ζητήσω από τον συνάδελφό μου από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ούτως ώστε να μιλήσει για την απλούστευση των προγραμμάτων. Αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι μια εργασία που κάνουμε από κοινού μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ενώ εξετάζουμε τις νέες πολιτικές για την ανακοίνωση για την, τον μηχανισμό ε, πολιτικής γειτονίας. Θα δώσω λοιπόν την, ε, το λόγο στον συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την Μεσόγειο. Θα ήθελα να πω ότι για την ώρα δεν υπάρχει πρόθεση να χρηματοδοτήσουμε πρόσθετες ανάγκες για την Νότιο Μεσόγειο εις βάρος των ανατολικών χωρών της πολιτικής γειτονίας. Θα πρέπει βεβαίως να, ε, να καταβληθούν πρόσθετες προστάσεις. Έχουμε όμως ευρύτερα θέματα τα οποία μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέσα του κεφαλαίου 4 ούτως ώστε να έχουμε πρόσθετα κίνητρα για τις χώρες της Νοτιού Μεσογείου με την αρχή more for more και με περισσότερη ερεσιμότητα και προαπαιτούμενα για να μην χαθεί αυτή η προσπάθεια έχουμε άλλες επιλογές στο κεφάλαιο 4 και δεν πρέπει να προσπαθούμε να αλλάξουμε τις, ε, τα κονδύλια που έχουμε, τις χρήσεις των κονδυλίων από την Ανατολή ε, προς τον Νότο από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, Διπλωματική Υπηρεσία. Καλημέρα σα Πρώτα να επιβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε πραγματικά εκ του σύνεγγυς με την ΤΕΦΚΟ για την ανάπτυξη. Η εκκίνηση τη διπλωματική υπηρεσία. δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι αυτό είναι ένα εμπόδιο στην ε, ακόμα περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μας που είναι εξαιρετική. Αυτό ήθελα να πω δεύτερον. Επιτρέψτε μου επίσης ε, σύντομα να θέσω στην ευρύτερη εικόνα της συζητή τι γίνεται σε σχέση με την περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι αυτή η εμπλοκή με τον Νότιο Καύκασο είναι ένα νέο σχετικά εγχείρημα. Ξεκινήσαμε μεγαλύτερη εμπλοκή με αυτές τις χώρες από το 2004, από την εκκίνηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Και στη συνέχεια ύστερα ξεκινήσαμε νέες διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Έχουμε μια συνεχή διαδικασία από το 2004 αναβάθμισης των σχέσεών μας. Το 2007 ήταν σχετικά πρώιμο σημείο στην διαδικασία αυτή τρία χρόνια μετά το 2004. Και θα ήθελα να πω ότι μόνο από το 2007 έχουμε πλήρως στελεχωμένες αντιπροσωπείες στην, στην Αρμενία και στην Γεωργία επίσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον προγραμματισμό, διότι πραγματικά οι αντιπροσωπείες μας είναι εκείνες που μας ενημερώνουν και μας εμπλέκουν στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Τώρα, να στραφώ στο θέμα ακριβώς το οποίο ζητήθηκε να τοποθετηθούμε. Ποια είναι τα μαθήματα που έχουμε συναγάγει από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα όσον αφορά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό. Θα ήθελα να αντανακλάτε σαφώς ότι ως αποτέλεσμα της ε, επανεξέτασης της πολιτικής γειτονίας και αυτό δεν είναι πια μυστικό για κανέναν θα υπάρξει μια πρόταση που θα εντάσει αυτές τις πτυχές στον προγραμματισμό μας ε, ήδη στο υψηλότερο επίπεδο διότι όπως αναφέρθηκε έχουν διαφορετικές φάσεις, διαφορετικά στάδια αυτά τα προγράμματα και θέλουμε πραγματικά να πλουστεύσουμε αυτή την προσέγγιση μας. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε, ή μάλλον να υπενθυμίσω κάτι. Έχουμε τις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης ε, και συνεργασίας ε, που αποτελεί τη νομική βάση ως πλαίσιο και καθορίζει τι θέλουμε να πετύχουμε και σε ποια κατεύθυνση θα στοχεύει το έργο μας. Και με βάση αυτό συντάξαμε προγράμματα δράσης και αναφορά έγινε στο πρόγραμμα δράσης για τη γεωργία με πολλές προτεραιότητες όπως αναφέρθηκε. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα, α, το ε, σχεδιασμού μόνο. Είναι ένα πολιτικό έγγραφο. Καλύπτει όλο το φάσμα, το εύρος των θεμάτων στην γεωργία όπως ε, μεταξύ μιας ε, εταιρικής χώρας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ολόκληρο εύρος φάσμα θεμάτων που θέλουν εκείνοι, αυτές οι χώρες δηλαδή, να προαχθούν. Και αυτό αναφέρει το τι θέλουμε να κάνουμε με μια τέτοια χώρα εταίρο, με βάση ακριβώς ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και στη συνέχεια η στρατηγική για τη χώρα και το, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, National Indicative Programs, καταδεικνύουν πώς συμπληρωματικά μπορούμε να δράσουμε, όπως στο επίπεδο τώρα της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης μπορούμε να συμπληρώσουμε. Έχουμε αρκετά έγγραφα. Δεν είναι όμως όλα προγραμματισμού έγγραφα, να μην υπάρχει παρανόηση από αυτού, είναι πολιτικής κατεύθυνσης έγγραφα. Και δεύτερον, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει χώρος για ευθυγράμμιση εδώ και απλούστευση και ένας από τους στόχους για την επανεξέταση, την αναθεώρηση θα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε και να εντάξουμε αυτές τις πτυχές ώστε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, να καλύψουμε ας το πω έτσι κάποια κενά και να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, να σα ρωτήσω, ικανοποιηθήκατε με αυτέ τι απαντήσει που πήρατε. Αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, να επανέλθω. Πάντα όταν γίνονται ενδιαφέροντα τα πράγματα σταματούν εκεί. Skip a step λέει. Να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Μέχρι πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα θέλω να ρωτήσω. Ακριβώς αυτό είναι το νευραλγικό σημείο όπου γίνονται τα πράγματα πιο εξειδικευμένα και είναι πιο ενδιαφέροντα. Τι θα γίνει λοιπόν. I Μπορώ να σας ζητήσω να απαντήσετε κύριε. Ξέρετε, αυτοί, αυτά τα αποτελέσματα της αναθεώρησης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα. Θα δημοσιοποιηθούν σε λίγες μέρες, σε κάποιες μέρες. Και από πλευρά των αρμοδίων θα δημοσιοποιηθούν. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Δεν μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι μπορείτε να αντιληφθείτε. Απλά και μόνο να σας πω ότι μας φαίνεται ότι θεωρούμε ότι πραγματικά μπορούμε να καλύψουμε ε, κάποια βήματα, κάποιες ενδιάμεσες φάσεις, να διασφαλιστεί η διατήρηση ενός μέσου, ενός εργαλείου που με βάση αυτή την εταιρική συνεργατική σχέση θα ταυτοποιήσουμε, θα εντοπίσουμε τα κύρια θέματα στα οποία θα εργαστούμε και με βάση αυτό θα υπάρξει ένα ενιαίο πρόγραμμα, ε, έγγραφο προγραμματισμού. Single programming, ε, programming document. Λοιπόν, ως η ερώτηση ήταν πότε θα μπορέσετε, όταν θα μπορέσετε να δημοσιοποιήσετε αυτά τα πράγματα, να δοθεί προσοχή σε αυτό το θέμα και έγκαιρα να μας ειδοποιήσετε. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Κύριε Ντεβρίς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χωρίς να επιθυμώ με κανένα τρόπο να ε, ακολουθήσω αυτές τις τόσο θελκτικές συζητήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ποια βήματα θα μπορούσαν να διαγραφούν ή να συνμηθούν από αυτό το μεγάλο μακρύ κατάλογο σε σχέση με τα θέματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου ένα θέμα είναι ότι τα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα θα μπορούσαν να εξεταστούν ως ένα από τα ενδυνάμει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να διαγραφούν. Όμως αυτό δεν θα έλυνε το μείζον πρόβλημα. Το κύριο θέμα είναι θα είχε νόημα για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον να εμπλακούμε σε μια σχετικά εκτενή συζήτηση με τις χώρες αποδέκτες για θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, για θέματα στρατηγικής, για κοινούς, αρκετούς κοινούς στόχους, joint objectives και μετά να περάσουμε στη συνέχεια σε μια δεύτερη φάση όπου θα δίνονται κονδύλια και να λαμβάνονται εκεί υπόψη θέματα τα οποία θα αποφασίζονται από εμάς τα οποία δεν βασίζονται υποχρεωτικά σε μια κοινή εκτίμηση. Το θέτω κάπως ε, σε αντίστοιξη μαύρο-άσπρο αυτό για να καταστεί πιο κατανοητό. Αυτό στο οποίο αναφέρομαι είναι η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δαπανώνται 50 έως 70% στον τομέα της δημοσιονομικής συνδρομής. Ακόμα και όταν χώρες αποδέκτες έχουν δείξει, έχουν επισημάνει ότι αυτά δεν θα ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα. Ο κίνδυνος είναι όσα περισσότερα εντάσσεται στη δημοσιονομική συνδρομή, τόσα λιγότερα θα βρίσκονται διαθέσιμα ως κονδύλια για χρηματοδότηση άλλων αναγκών. Και σε σχέση με το Αζερμπαϊτζάν για την περίοδο προγραμματισμού ελήφθησαν υπόψη τέσσερις από τις δέκα υποπροτεραιότητες. Αυτό είναι θέμα Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποφασίζεται, δηλαδή για τις επιλογές που θα γίνονται. Και αυτό έχει συγκεκριμένες ε, επιπτώσεις, συγκεκριμένες συνέπειες. Είναι σημαντικό αυτό να γίνει αντιληπτό. αντιληπτό. Να μην υπάρξει παρανόηση, αλλά σε σχέση με τη χρήση του όρου διαφθορά, ελπίζω ότι κατέστησα σαφές ότι αυτό δεν είναι σε σχέση με την χώρα την οποία συζητούμε με τις χώρες που συζητούμε, αλλά είναι υπό το πρίσμα των γενικότερων συζητήσεων που διεξήχθησαν εχθές για την δημοσιονομική σύνδρομη. Θα πρέπει να αντανακλάται εδώ το μέλημα ότι η γενική σύνδρομη δεν βασίζεται πάντα σε επαρκή, ε, σε επαρκή εχέγγυα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αυτό πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσει στο να προσέξουμε περισσότερο αυτά τα θέματα στην ε, καθημερινή δουλειά. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν σε αυτό το τμήμα. Σημείο 18 της ημερήσιας διάταξής μας σήμερα είναι τα διάφορα. Υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να θίξει κάτι υπό τα διάφορα. Όχι. Έχουμε ημερομηνίε των επόμενων συνεδριάσεων. Είναι γνωστές σε όλους μας να υπενθυμίσω 24 και 25 Μαΐου 2011. Σας ευχαριστώ όλους σας. Καλό σας ε, γεύμα. Καλή όρεξη. Γεια.